Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 like eh, eh, <laughs> at Παρακαλώ, καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας και έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς και από. Παρακαλώ ελέγξτε τα ακουστικά σας για να μπορέσετε να ακούσετε. Ehm, λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω σήμερα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Γιάσικ Μπούζεκ, ο οποίος ε, θα προεδρεύσει τις ενακτήρια συνεδρίασης ε, αυτής της ε, διάσκεψης. Σας καλωσορίζω κύριε Πρόεδρε και σας δίνω αμέσως το λόγο. Τι καλά που μαθαίνουμε γλώσσες, λέει ο πρόεδρος του σώματος και έτσι μπόρεσα να σας καταλάβω κυρία πρόεδρε, χωρίς να χρησιμοποιήσω τα ακουστικά μου. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη και αγαπητοί εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Σήμερα γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα των γυναικών και επιλέξηκε πιστεύω το καλύτερο θέμα για αυτήν την ε, συνεδρίαση η βία κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών, που είναι μια θλιβερή πραγματικότητα στον κόσμο. Πρέπει να αρχίσουμε να καταπολεμούμε αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο να το συζητάμε. Το Ευρωμεσογειακό, η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση υιοθέτησε μία σύσταση και στην Ολομέλεια όπου κάλυψε πάρα πολλά σημαντικά σημεία τον ε, μοναδικό ρόλο των γυναικών, την ε, υλοποίηση μέτω για την προστασία των γυναικών, τον σεβασμό της αξιοπρέπειας, ε, την ενίσχυση στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των γυναικών και άλλα παρόμοια σημαντικά μέτρα και συστάσεις. Βεβαίως δεν έχουμε μόνο κατά νου τη Μεσόγειο, και την ε, Ανατολική Δυτική Μεσόγειο και τις ε, χώρες αυτές της ε, Νότιας Ευρώπης. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες τις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επιτροπή Γυναικείων Υποθέσεων και όλους τους διοργανωτές αυτές της της, της διάσκεψης που οργάνωσαν αυτήν την ακρόαση και επίσης το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, το Συμβούλιο Ευρωπαίων Καταναλωτών και όλες τις συναφείς οργανώσεις που συνέβαλαν και το ΕΦΣΚΟ έχει οργανώσει ε, στα πλαίσια του ΟΗΕ και το, ε, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη έχει οργανώσει παρόμοιες ε, διασκέψεις και συνέδρια για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών κύριε Πρόεδρε, μια που έχουμε την θαυμάσια δυνατότητα διερμηνίας σε όλες τις γλώσσες, θα συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα που είναι τα πολωνικά. Ξέρουμε τα στατιστικά στοιχεία ότι 15% των γυναικών στην Ευρώπη έχουν ε, υπάρξει θύματα βίας και μάλιστα σε καθημερινό επίπεδο. Η βία κατά των γυναικών είναι ε, ποινικό αδίκημα όχι μόνο κατά του ατόμου αλλά και κατά της ανθρωπότητας. Έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητος και δεδομένου ότι αυτό το θέμα θίγει το ίμιση των Ευρωπαίων πολιτών, θεωρούμε το ψήφισμα το οποίο ε, εκδόθηκε πέρσι τον Εύριο για τη βία, η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα του σώματος. Δεν είναι καινούριο θέμα αυτό, αλλά αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε στις, να ενισχύσουμε τη βοήθεια που προσφέρεται σε αυτές τις γυναίκες, να ξεπεράσουν τις φοβίες, να ξεπεράσουν τον τρόμο να ξεπεράσουν το αίσθημα της ε, απελπισίας ε, και ε, το ότι είναι αβοήθητες και δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει και να τις προστατεύσει. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να κατηγορήσουν πολλές φορές και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους ε, ανθρώπους που ε, διαπράττουν αυτά τα δικήματα βίας, οι οποίοι συνήθως είναι άνθρωποι του στενού και ονιακού περιβάλλοντος, είναι μέλη της οικογένειάς τους, οι σύντροφοι και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και την Ισπανική Προεδρία, η οποία είχε ε, βάλει το θέμα αυτό ως θέμα προτεραιότητος στην ατζέντα. Είχα επισκεφθεί μαζί με τους εκπρόσωπους της Ισπανικής κυβέρνησης ένα συνέδριο που είχε γίνει επί Ισπανικής Προεδρίας και είχαμε συζητήσει πολύ αυτό το θέμα και επίσης στο Ευρωπαϊκό ε, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Το θέμα αυτό παρακολουθείται στενά και η εξέλιξη όλων των συναφών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ και την αρμόδια επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ. Η Europol δεν ασχολείται με το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Δεν υπάρχουν ε, στατιστικές, ε, στατιστικά προγράμματα ούτε προγράμματα πρόληψης. Αυτό το διαπίστωσα πριν από μερικές μέρες όταν έψαχνα το διαδίκτυο για πληροφορίες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και στην εργασία τους, διότι δεν την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισης όπως οι άνδρες. Επίσης αυτό φαίνεται ιδιαίτερα τώρα σε περίοδο υψηλής ανεργίας. Ένα άλλο θέμα είναι βεβαίως η εξισορρόπηση της ε, εργασίας με την οικογενειακή ζωή. Οι μητέρες πρέπει να ενισχύονται, πρέπει να υπάρχουν μέτρα υποστήριξης για να μπορέσουν να συμφιλιώσουν την οικογενειακή με την εργασιακή ζωή. Πρέπει να δώσουμε οικονομικά κίνητρα, πρέπει να ε, δημιουργήσουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει την ε, ελαφρύτερη φορολόγηση όταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά στην οικογένεια πολύ τεχνικό γένεια, λιγότεροι φόροι. Σήμερα είναι παρόντες μαζί μας πολλοί κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από άλλες χώρες και είναι σε πολλές χώρες δραματικά τα στοιχεία της βίας κατά των γυναικών. Ιδίως η βία ε, κατοίκων, η οικογενειακή βία. Θα ήθελα να, δια, διαβεβαιώσω όλα τα μέλη και όλους τους παρόντες ότι έχω προσωπικά δεσμευτεί να ε, κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημα μπορούμε να τη σταματήσουμε, μπορούμε να τη σταματήσουμε τη βία. Είναι ένα πλήγμα κατά της κοινωνίας. Δεν είναι μια κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζούμε. Μια κοινωνία που, που έχει βία κατά των γυναικών, όπου σημειώνεται βία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι με, μεγάλη χαρά ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Σώματος, τον κύριο Μπούζεκ, για την ε, εξαιρετική του εισήγηση σήμερα και για την θαυμάσια εργασία την οποία έχει επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την Προεδρία του. Έχει πραγματικά δεσμευτεί έντονα και εις βάθος στο θέμα αυτό και σε όλα τα γυναικεία θέματα. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα ε, τον Πρόεδρο κύριο Μπούζεκ. Επίσης με μεγάλη χαρά καλωσορίζω σήμερα τα μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου και ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως ε, όλους τους συμμετέχοντες και ομιλητές ε, και ομιλήτριες. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω επίσης και να καλωσορίσω τους πολίτες που είναι εδώ παρόντες από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολίτες οι οποίοι έχουν συμβάλει σε αυτήν την εκστρατεία, έχουν σχεδιάσει ε, την αφίσα, το πόστερ αυτό που βλέπετε με το σύνθημα Καλωσορίσατε λοιπόν στην συνεδρίασή μας αυτή. Οι τρεις, αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι, ήταν υπεύθυνοι για την, τον σχεδιασμό και την προβολή αυτού του πόστερ. Μαζί με την ε, Διεθνή ημέρα της γυναίκας και παράλληλα με αυτήν την ε, ευκαιρία μπορέσαμε να ανταλλάξουμε πάρα πολλές απόψεις και να ενημερωθούμε για το τι γίνεται διεθνώς σε παρόμοια θέματα. Εκτός μικροφώνου, κόπηκε το μικρόφωνο της Πρόεδρου ξαφνικά και χάσαμε τον ήχο. Εντάξει. Το θέμα το οποίο διαλέξαμε σήμερα, βία κατά των, ε, φέτος, ε, βία κατά των γυναικών, είναι ένα ευρύτατο πρόβλημα και εκφράζεται με διαφορετικές μορφές. Βασίζεται κυρίως σε, στο θέμα του φίλου Είναι βία εναντίον ενός συγκεκριμένου φίλου κατά συντριπτική πλειοψηφία. Βεβαίως, Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ισπανική Προεδρία που έθεσε το θέμα αυτό στον ε, κατάλογο προτεραιοτήτων διότι πάντοτε πιστεύαμε ότι είναι ένα ε, πολύ ε, σημαντικό πρόβλημα και ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει, να βρούμε τρόπο να σταματήσει αυτή η βία. Γι' αυτό ακριβώς επιλέξαμε και αυτό το μήνυμα. We can stop it. Μπορούμε να τη σταματήσουμε, τη βία ή να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι δυνατόν, μπορούμε. Σήμερα θα ακούσουμε διάφορους ομιλητές, εκπροσώπους από οργανώσεις που καλύπτουν και το θέμα της βίας κατά των γυναικών και είμαι βέβαιη ότι σήμερα θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις από τους ομιλητές μας και θα μας προβάλλουν ιδέες και προτάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εξάλληψη αυτού του φαινομένου της βίας. Υπάρχει πρόταση, ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 2010 ψήφισμα του σώματος. Η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ επίσης θα μας ενημερώσει για την εμπεριστατωμένη μελέτη την οποία έκανε η Κομισιόν με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας μεταξύ των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βία κατά των γυναικών είναι ένας ε, τομέας, ε, ένα θέμα υψίστης ε, προτεραιότητας όταν ρωτάμε τους πολίτες μας τι πιστεύετε ότι μπορούμε και τι και πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνέχεια. Γι' αυτό είναι πολύ θετικό βήμα για μας να αναπτύξουμε αυτή την πρωτοβουλία η οποία πραγματικά καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των ανησυχιών ε, και των ε, ενδιαφερόντων των πολιτών μας. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Υπουργό Ισότητος ε, της Ισπανίας, και δεδομένου ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί τόσο υψηλά στην ατζέντα, καλωσορίζω την κυρία Μπιβιάνα Αΐντο Αλμάγκρο, Υπουργό σε θέματα ισότητος ε, από την, της Ισπανίας, η οποία έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Προεδρείο, κυρίες και κύριοι, πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω διότι μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση της ε, Διεθνούς Μέρας της Γυναίκας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλους τους δημοκράτες πέραν από τις ευθύνε ε, και αρμοδίες που έχει ο καθένας είναι μια τιμή κανεί να μιλάει εδώ σε αυτό το εμικύκλιο του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί εκατομμύρια πολιτών της Ευρώπης των 27 κυρίες και κύριοι στην σημερινή συγκυρία έχουμε φτάσει σε μια στόχη πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τον 21ο αιώνα διότι αρδενώς έχουμε τώρα αυτή την εδραίωση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτούς τους κοινούς θεσμούς διότι με αυτόν τον τρόπο τώρα ε, έχουμε την αύξηση των δημοκρατήτων αυτού του κοινοβουλίου από την άλλη μεριά, έχουμε ένα προγραμματισμό πιο εδρεωμένο από την επόμενη δεκαετία ε, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την χρηματοπιστωτική διεθνή κρίση και έτσι να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Επομένως η σημερινή χρονιά θα είναι πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη για την ισότητα των γένων. Θα έχουμε έναν ε, στόχο ε, το οποίο δεν απεμπολούμε ποτέ για όλες τις πολιτικές που αναπτύσσουν τις επιμέρους και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για, το, για την υπόθεσή μας στον ΟΗΕ γιατί έχουμε 15 χρόνια που ισχύει η πλατφόρμα του Πεκίνου ε, και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε 17 κυβερνήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τον Φεβρουάριο στο Κάδες επιβεβαιώσαμε ότι θέλουμε να υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών στις ε, αποφάσεις τις ε, οικονομικές, τις πολιτικές και επιχειρηματικές στην Ευρώπη. Οπότε ε, σε αυτό το, το πλαίσιο ε, με αυτοκριτική, με δεσμεύσεις. Έχουμε καθορίσει αυτό το καινούργιο στόχο στην Ευρώπη, οπότε δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε την βία κατά των γυναικών. Και θα πρέπει να συγχαρώ το Κοινοβούλιο, γιατί πάρα πολύ σωστά ε, προχώρησε σε αυτή την ε, εκδήλωση και σε αυτή την πρωτοβουλία κατά της βίας κατά των γυναικών. Επομένως θα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε βία βασκείται κατά των γυναικών και θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε την, ε, την βία των που γίνεται στο σπίτι, αλλά θέλω να αναφέρω και το, το δουλεμπόριο ε, και η σεξουαλική εκμετάλλευση. Και αυτό είναι η πρόκληση για τον επόμενο αιώνα, για τον, για τον 21 πρώτο τον αιώνα μας στα πλαίσια του ΙΕ όπως κρίθηκε και υπάρχει βέβαια και, υπάρχουν και κάποιες εθνικές ε, παραδόσεις, πολιτικές παραδόσεις που είναι κατά των γυναικών όπως οι σεξουαλικοί ακροτηριασμοί η αναγκαστική γάμη και τα εγκλήματα τιμής. Οπότε όλα αυτά είναι εκδηλώσεις βίας και όλα αυτά κατατείνουν στην ανισότητα ανδρών και γυναικών. Έχουμε μια κουλτούρα κυριαρχής από των γυναικών, κάτι το οποίο περνάει μέσα από όλη την ιστορία σε όλες τις κοινωνίες. Είναι μια ιστορική τάση για την οποία είμαστε υπεύθυνοι ε, όσο γίνεται μέσα και έξω τα σύνορα γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στον πολιτισμό και στη δημοκρατία. Πρόκειται για βία κατά του μισού πληθυσμού της γης που ασκείται κατά ανθρώπων ιδιότι τυχαίνει να είναι γυναίκες. Τελευταία 15 ετία στην Ευρώπη μπορούμε να δούμε ότι έχουμε πετύχει κάποια πράγματα αλλά ακόμα κάποιοι άλλοι στόχοι εκκρεμούν όπως το να μπορέσουμε να σταματήσουμε τέτοιου είδους βία. Επομένως, είναι κάτι που ακόμα πρέπει να το κάνουν πολλά κρατή-μέλη, θα πρέπει να υπάρχουν εθνικά προγράμματα κατά της βίας μεταξύ των δύο φύλων. Θα πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί ε, το σχετικό έγκλημα στο ποινικό δίκαιο. Οπότε θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι έχει γίνει το 2010 ένα σημαντικό βήμα πρόοδο, διότι πριν από μια εβδομάδα οι Υπουργοί Απασχόληση Γενικής πολιτική και Κατανάλωσης ενέκριναν κάποια συμπεράσματα για τον αποκλεισμό της βίας κατά της γυναίκας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι οι 27 έβαλαν τι βάσεις για να υπάρχει ενιαία δράση στην Ευρώπη κατά τις δράσεις κατά γυναικών. Και με τις εξελίξεις για τη χάρτα των δικαιωμάτων και την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ο πολίτης είναι στο επίκεντρο των κοινοτικών πολιτικών. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που συζητούμε, το οποίο είναι καθημερινό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει σχέση με τους στόχους και τις φιλοδοξίες της Ευρώπης. Και η Ευρώπη έτσι θα αναδειχθεί όταν προστατεύει κάθε γυναίκα που είναι θύμα βίας ε, της ε, βίας κατά των γυναικών και να καταπολεμηθεί με θάρρος σε όλες τις μορφές της. Να γίνει δράση κοινή, με πρόληψη και επίσης να υπάρχει αρρωγή προς τα θύματα της βίας και ε, αυτά τα συμπεράσματα κατατείνουν σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για πρόληψη και καταπολέμηση της βίας. Και θα γίνει αυτό τη βάση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε έτσι να έχουμε μια πλατφόρμα που θα συγκεράζει τις εμπειρίες των κρατών μελών, των φορέων, των οργανώσεων γυναικών για να μπορούμε να αποκλείσουμε αυτού του είδους τη βία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να γίνει το ίδιο και έξω από τα σύνορα της Ένωσης και έτσι να έχουμε τελικά κάποια κριτήρια κοινά για τους 27, μεθοδολογία, συλλογή δεδομένων, όλα αυτά τα οποία περιέχει η έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά την αναδοχή της πλατφόρμας του Πεκίνου στην ε, Ένωση. Έτσι να χαράξουμε τις ε, πολιτικές μας και να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σχετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Γιατί έχει συμφωνηθεί ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ε, την συγκρότηση ενός παρατηρητηρίου ευρωπαϊκού για την βία των γυναικών. Μόνο με τη γνώση θα ξεπεράσουμε τους μύθους και θα φτάσουμε στη γνώση μέσα από τη συλλογή των πληροφοριών. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μελέτη, παρατήρηση αλλά και δράση. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης που να είναι συνεχής για πρόληψη, επισήμανση, για τέτοιου είδους στερεότυπες συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε άσκηση βίας. Επομένως πρόκειται για έργο πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά ιδίως τους νεότερους. Επομένως έτσι θα πρέπει να προβάλλουμε το πρόβλημα για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά. Αυτό το οποίο γίνεται ενίκο να ξεμπροστιαστεί, να γίνει δημόσια υπόθεση και να γίνει ευθύνη όλης της κοινωνίας. Άρα, έτσι θα έχουμε ως στόχο την συνειδητοποίηση στην Ευρώπη του ότι θα έχουμε ε, φέτος αυτό το, ή κάποια στιγμή την χρονιά αφιερωμένη στην κατανόηση της βίας. Επίσης, να έχουν τα κρατη τα μέσα για να βοηθούν τα θύματα, όπως έναν αριθμό τηλεφώνου που μπορεί κανείς δωρεάν να τηλεφωνήσει, όπως το 116 το οποίο έχει θεσπιστεί ήδη να σταματήσουν οι γυναίκες να υφίστανται αυτή τη ε, βία σε όλες τις ε, εκδηλώσεις της ζωής. Έχουμε επίσης και ένα σχέδιο οδηγίας για προστασία της γυναίκας. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην περίπτωση που έχουμε θύματα διαφόρων εγκλημάτων μεταξύ των οποίων και τα εγκλήματα μεταξύ των δύο φύλων. Οπότε θα πρέπει να μπορούν να ασκήσουν το θεμητό του δικαίωμα οι γυναίκες να είναι προστατευμένες, να μην καταλήγουν σκλάβοι, δούλοι, καμία. Ούτε από φόβο, ούτε από αυτά τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων. Γιατί είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και δεν θέλουμε να γίνεται αυτό το πίγνι και στην, στην ελληνική μυθολογία με την απαγωγή της Ευρώπης. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η δέσμευση της Κομισιόν ούτω ώστε να προχωρήσει μία οδηγία αυτό το εξάμεινο κατά αυτή την Προεδρία κατά της διακίνησης γυναικών για λόγους εξχολής εκμετάλλευσης. Οπότε να έχουμε τελικά μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την βία κατά των γυναικών. Να σταματήσει αυτό να είναι καθημερινή πραγματικότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Να μην είναι κάτι το οποίο το αποδεχόμαστε, κάτι στο οποίο ε, αδρανούμε και έτσι έμεσα συνενούμε. Να είναι κοινό στόχος αυτό να μπει στην πολιτική μας ατζέντα και να προχωρήσουμε σε κάποια οδηγία είπαμε ή σε κάποια συμπεράσματα, κάτι το οποίο έγινε και αυτό είναι μόνο μια αφετηρία για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την βία, να αποκτήσουμε την, ε, μια κουλτούρα που να αντιβαίνει σε αυτή την ε, ε στην, στην βία και όπως είπαμε και στις 11 Μαρτίου μπορούμε να σταματήσουμε τη βία των γυναικών αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε σε προσπάθειες γιατί είμαστε σε μια εποχή αλλαγών, αλλά οι αλλαγέ δεν γίνονται από μόνε του. Και γι' αυτό το λόγο η συνεργασία του Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα οδηγήσει ε, σε κάποια αποτελέσματα που και αυτό είναι συνθήκη εκ των ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό τον σημαντικό στόχο. Ενωμένοι να καταπολεμήσουμε την βία για τα δικαιώματα των θυμάτων με πρόληψη, με ε, εκπαίδευση και έτσι να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κυρία Ιντο Αλμάγκρο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο και η, προεδρία, η ασκούσα Προεδρία του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση ακριβώς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα με μεγάλη μου χαρά να καλωσορίσω την Αντιπρόεδρο της ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ε, κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ, που είναι υπεύθυνη για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των πολιτών. Ένα θερμό καλώς όρισμα λοιπόν από εμάς, ε, κυρία Ρέντινγκ, και έχετε ευθύς αμέσως το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί βουλευτές, και κύριοι, γιατί πέρα από τις κυρίες υπάρχουν και κάποιοι κύριοι από το σώμα. Να τους καλωσορίσουμε λοιπόν θερμά, διότι θέλουμε τη βοήθειά τους. Θέλουμε να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μπορέσουμε μαζί να γιορτάσουμε την Διεθνή Μέρα της γυναίκας από την 8η Μαρτίου. Βέβαια έχουμε ξεπεράσει κατά κάποιες ημέρες την 8η Μαρτίου, αλλά αυτό δεν πειράζει, διότι νομίζω ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι μέρα της γυναίκας. Κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας εδώ και 100 χρόνια που γιορτάσαμε την πρώτη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας για πρώτη φορά και έχουμε καταφέρει πολλά έκτοτε. Όμως ακόμη ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς κατά κύριο λόγο ε, σε σχέση με το σημερινό μας θέμα, την βία κατά των γυναικών. Κάτι που δείχνει πόσο σοβαρές είναι οι προκλήσεις που έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Είναι μεγάλη μου η ευγνωμοσύνη μου προς τους διάφορους ε, υποστηρικτές της διοργάνωσης της σημερινής είναι μεγάλη και επίσης προς την Προεδρία την Ισπανική, η οποία περιέλαβε την ε, βία κατά των γυναικών ως ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα μεταξύ των προτεραιοτήτων της. Στις 5 Μαρτίου, λίγες μέρες πριν την ε, Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, ο πρόεδρος Μπαρόζο και εγώ ίδια, ένας άνδρας και μια γυναίκα, παρουσιάσαμε από κοινού την χάρτα για τις γυναίκες. Η χάρτα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν είναι απλώς μια πολιτική δήλωση του κολεγίου των 27 επιτρόπων είναι επίσης μία δέσμευση των 27 επιτρόπων να εφαρμόσουν τα θέματα ισότητας των φύλων και να τα ενσωματώσουν σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα ρεκόρ. Είναι μία πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή έχει εγκρίνει αυτή τη χάρτα και όλοι οι επίτροποι θα συνεργαστούν προκειμένου η διάσταση για τα δύο φύλλα και ορατή να είναι και να ενσωματώνεται σε κάθε μια πολιτική μας ξεχωριστά. Η χάρτα εντοπίζει πέντε τομείς κλειδιά για τη δράση μας τα ερχόμενα πέντε χρόνια. Ένας από αυτούς τους τομείς δράσης ονομάζεται αξιοπρέπεια, ακαιρεότητα και να δοθεί τέρμα στην βία ε, που ασκείται μεταξύ των δύο φύλων. Διότι γνωρίζουμε ότι κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχει ακριβώς να κάνει με τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα των συνθήκων μας. Θα πρέπει λοιπόν η χάρτα αυτή να λειτουργήσει. Αυτή είναι η πηξίδα μας. είναι αυτό που θα μα οδηγήσει στην πορεία μα. Και όλε μα οι δράσει πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με αυτή τη χάρτα. Είδαμε ήδη σήμερα ότι ό,τι έχει να κάνει με την βία δεν είναι θέματα που πρέπει να τα συζητάμε μόνο εδώ στι Βρυξέλλε που χτίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχουμε έρθει σε επαφή με γυναίκε όλη τη Ευρώπη μέσω του Ευρωβαρόμετρου. Ναι, λοιπόν, δεν υπήρξε ούτε μία εξαίρεση. Όλε οι Ευρωπαίε γυναίκε πιστεύουν ότι η βία είναι το νούμερο ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έκανε τη σωστή επιλογή. Η βία είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να εξαλειφθεί η βία. Εκφράζω λοιπόν την ευγνωσύνη μου και προς την κυρία Σβένσον, η οποία προσωπικά μίλησε για το τεράστιο προσωπικό κόστος της βίας στη δική της οικογένεια και μας είπε και εδώ αναφέρω τα λόγια της, να φανταστούμε κάθε στιγμή της ζωής μας να φοβόμαστε τον σύντροφό μας, τον άνθρωπο με τον οποίο έχει κανείς σχέση. Ε, διότι τον κατηγορούμε συνεχώς και βεβαίως εκείνος ελέγχει τα πάντα. Είναι λοιπόν σημαντικό οι γυναίκες επιτέλους να μιλήσουν, να λάβουν το λόγο, διότι πολύ συχνά αυτό το είδους ιδέα παραμένει ταμπού. Πρέπει λοιπόν αυτό το ταμπού να το πολεμήσουμε Πραγματικά ε, ενθαρρύνω όλες τις γυναίκες της Ευρώπης να πάρουν το λόγο και να μιλήσουν για αυτό το ταμπού, να υψώσουν τη φωνή τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο επίπεδο της οικογένειας και του οικογενειακού βίου. Υπολογίζουμε ότι το 1 πέμπτο ή το 1 τέταρτο των γυναικών της Ευρώπης έχουν αντιμετωπίσει μορφές βίας κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους και 1 τρίτο επίσης έχουν ε, και μάλλον ένα μικρότερο ποσοστό έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Ξέρουμε ότι πολλές γυναίκες ζουν σε ακόμη χειρότερες συνθήκες και Είμαστε ευγνώμονες προ την Επίτροπο, την κυρία Μάλστρομ, ειδική επιτετραμένη των Ηνωμένων Εθνών, για την παρακολούθηση και τη μέρημνα επί των γυναικών σε συνθήκες πολέμου. Εδώ άκουσα την εκτίμησή σας ότι περίπου 500.000 γυναίκες που ζουν στην Ευρώπη έχουν υποφέρει την, ε, τον γυναικείο εκοτεριασμό των σεξουαλικών οργάνων. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι καθημερινά 600.000 κοπέλες παγκοσμίω είναι θύματα βασαναστηρίων αυτό είναι ένα φρικτό έγκλημα. Ούτε μπορεί να το αποδεχόμαστε. Ούτε στην Ευρώπη ούτε πουθενά στον κόσμο. Διότι η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το αίτιο των ε, ηθών, των παραδόσεων, των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Είναι έγκλημα τελεία. Και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε όλα αυτά να πάυσουν. Η Επιτροπή λοιπόν επιβεβαιώνει τη σοβαρή τη δέσμευση να καταπολεμήσει τη βία κατά των γυναικών. Η δέσμευσή μα πρόκειται να αντικατοπριστεί στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, κυρίω των γυναικών που είναι θύματα βία και του ακροτηριασμού των γενετικών οργάνων. Η κυρία Μάλστρομ και εγώ ίδια σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα δράση που θα παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό και θα φροντίζει να ε, περιγράφει την υλοποίησή του. Η βία και η, η παρακολούθηση των ε, θυμάτων της βίας θα είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Τις ερχόμενες, τις ερχόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε με προτάσεις για, ποινικό, για να περιληφθούν σε κώδικες ποινικού δικαίου και να καταπολεμηθεί με τον τρόπο αυτό η εμπορία ανθρώπων. Επίσης θα ενισχύσουμε το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο εδώ και μια δεκαετία παρέχει στήριξη σε δράσεις για την καταπολέμηση βίας κατά των παιδιών, νεαρών ανθρώπων και γυναικών. Θα προστατεύσουμε θύματα και ομάδες που απειλούνται. Ως τώρα το πρόγραμμα Δάφνη έχει χρηματοδοτήσει 500 προγράμματα τουλάχιστον. Βλέπετε λοιπόν, Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δραστηριοποιηθεί εντατικά ω τώρα για τα θέματα αυτά. Στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη ξεκινήσαμε και μία μελέτη για τις βλαβερές παραδοσιακές ε, πρακτικές. Ανέφερε κάποιες υπουργό τους κατά εξαναγκασμού γάμους ή τον ε, γυναικείο ακροτεριασμό των ε, γεννητικών οργάνων. Τον Απρίλιο θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και το πόρισμα αυτό θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε δράσεις προκειμένου να πάυσουμε τον γυναικείο εκοτριασμό βασισμένοι σε αποδεδειγμένες και ελεγμένες πρακτικές από την Ευρώπη και αλλού και στην νομοθεσία και στη χάραξη πολιτικών και στην πράξη και συμπεριλαμβάνοντας τη συνεργασία μας με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν βοηθήσει δηλαδή τις γυναίκες που ήταν θύματα ακροτεριασμού. Επίσης θα ήθελα να εντατικοποιηθεί η δράση μας για την βία που, τα φαινόμενα βίας μεταξύ των δύο φύλων και Βεβαίω για να πάυσουν οι περιπτώσεις, να εξελιχθούν όλες οι περιπτώσεις ε, του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποινικά μέτρα όπου χρειάζεται. Καλέστε την Επιτροπή να σκεφτεί μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση της νομοθεσίας για θέματα αυτά. Για τη βία, τα φαινόμενα βίας μεταξύ των δύο φύλων και κατά των παιδιών μην ξεχνάμε ότι στα παιδιά συμπεριλαμβάνονται και τα νεαρά κορίτσια. Αλλά κάποιε φορέ έχουμε φαινόμενα βία και κατά των ε, μικρών αγοριών. Περιμένω τα πορίσματα τη μελέτη μα λοιπόν να μα δείξουν δυνατότητε για εναρμόνιση τη νομοθεσία μα. Πρόεδρε, τον Νοέμβριο πέρυσι σε αυτό το σώμα ζητήσατε μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική προκειμένου να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές βίας Νωρίτερα τον ε, τρέχοντα μήνα, το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Ιδού η απόκρισή μου. Τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια συνολική στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών που θα καλύπτει την περίοδο 2010-2015. Η στρατηγική αυτή θα μετατραπεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι καθοριστικές αρχές που ανακοινώνονται στην χάρτα για τις γυναίκες καλύπτει ως γενική οδηγητική γραμμή την, το πλαίσιο αυτό της Επιτροπής. Και εδώ θα καλύπτουμε και πολύ συγκεκριμένους τομείς. Επίση, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να οργανώσει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου, Πρόεδρε, προκειμένου να διαμορφώσουμε συνεκτικότερε πολιτικέ που να ασχολούνται με όλα τα φαινόμενα βία κατά των γυναικών. Εδώ, με μεγάλη μου χαρά, μπορώ να σα επιβεβαιώσω ότι θα διοργανωθεί η διάσκεψη αυτή στι 25 Νοεμβρίου φέτο, προκειμένου να γιορτάσουμε τη Διεθνή ημέρα εξάλληψη τη βία κατά των γυναικών. Αυτή η ευκαιρία θα μα επιτρέψει να παρουσιάσουμε τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και βεβαίω θα είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και του ενδιαφερόμενου, του συμμετέχοντε, τι εθνικέ κυβερνήσει, τα εθνικά κοινοβούλια και τα μέλη τη κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση εξακολουθεί τι διαπραγματεύσει τη στο Συμβούλιο τη Ευρώπη για την Σύμβαση πρόληψη και Καταπολέμησης τη βία κατά των Γυναικών και το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων θα τροφοδοτήσει το έργο μας. Βλέπετε λοιπόν, Πρόεδρε, ότι το πράγμα αυτό μας απασχολεί σοβαρά. Η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα. Έτσι να την αποκαλούμε. Και ας το πούμε και στον κόσμο, ανοιχτά είναι έγκλημα. Βεβαίω, εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όπως λέει και το σύνθημά σα, μπορούμε να την αναχαιτήσουμε αυτή τη βία. Αλλά είμαι πεπισμένη, Πρόεδρε, ότι αν θέλουμε να τα καταφέρουμε, όχι μόνο μπορούμε να εξαλείψουμε τη βία, αλλά θα τα καταφέρουμε, θα την εξαλείψουμε. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ρέντιν για την εμπνευσμένη της αυτή ομιλία. Θέλουμε η άριστη αυτή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχιστεί. Όπως είπε η Επίτροπος Ρέντινγκ στην αρχή της παρέμβασής της, θα αντλήσουμε διδάγματα από τις εμπειρίες που ήδη έχουμε και θα αξιοποιήσουμε όλες τις εμπειρίες που μπορούν να μας παράσχουν με κυβερνητικέ οργανώσεις και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πεδίο αυτό. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν την παραμικρή γνώση και εμπειρία που μπορεί να διαθέτουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερος. Ευχαριστούμε και την Υπουργό για τα θέματα ισότητας από την Ισπανία, την κυρία Αίντο Αλμάγκρο και την Επίτροπο Ρέντινγκ. Και τέλος να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μπούζεκ, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, για την εμπνευσμένη του επίσης ε, παρέμβαση στην αρχή της σημερινής συζήτησης. Ξεκινάει τώρα η αυτή καθ' αυτή συζήτηση. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι θα πρέπει να έχετε βρει ένα έντυπο στα έδρανα μπροστά σας. Και αν θέλετε να λάβετε το λόγο, θα πρέπει να το έχετε συμπληρώσει. Μπορούμε να επιτρέψουμε ένα δίλεπτο ομιλία σε κάθε παρεμβαίνοντα. Θα είναι σημαντικό λοιπόν ο καθένας να περιοριστεί στο χρόνο αυτό ομιλίας για λόγους ευγένειας και σεβασμού, και να ακούσουμε και όσο το δυνατόν περισσότερους ομιλητές βεβαίως. Είστε λοιπόν ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στη συζήτηση και απλώς ε, μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο αν θέλετε να μπορέσετε να λάβετε το λόγο. Και τώρα να δώσω το λόγο στους πρώτο, στον πρώτο από τους ομιλητές μας, στην πρώτη από τις ομιλητριές μας μάλλον, την κυρία Μητρία από την ε, Ρουμανική Γερουσία. Έχετε το λόγο. Η κυρία Μητρέα. Ναι. Και περιμένουμε την κυρία Μητρέα. Οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Ματέρα εντωμεταξύ. Ζητώ συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Η κυρία Μητρέα δεν είναι εδώ ακόμα. Έχουμε αυτό τον μακρύ κατάλογο μιλωτών. Α, καταρχάς λοιπόν η Βαρόν Βίτμαρ από τη Βουλή των Λόρδων στον Ηνωμένο Βασίλειο. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Στη Μεγάλη Βρετανία μία από τις τέσσερις γυναίκες είναι θύματα οικιακής βίας όμως έχουμε πολιτιστικές ε, ιδιαιτερότητες, δεδομένου ότι είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Προέρχομαι εγώ από ένα πολιτιστικό περιβάλλον όπου η βία στο σπίτι θεωρείται έθιμο, παράδοση. Και πρέπει να πω ότι η κοινωνία των πολιτών φοβάται να καταγγείλει τις ε, πολιτιστικές, ε, τα πολιτιστικά δικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις γυναίκες, ιδίως σε αυτές τις κοινότητες όπου η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη και όπου η γυναικεία φωνή δεν ακούγεται, διότι πολλές φορές οι γυναίκες είναι σήματα, αλλά κρύβονται, δεν ακούγονται, δεν φαίνονται Το θέμα είναι να έρθουμε σε επαφή με τις χώρες και τα κοινοβούλια των χωρών της προέλευσης των γυναικών αυτών που προέρχονται από πολιτιστικές μειονότητες και να διαβουλευτούμε με τα κοινοβούλια και τους εθνικούς αντιπροσώπους να δούμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Το πρόβλημα αυξάνεται, μεγαλώνει, δεν ε, περιορίζεται. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ματέρα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν μεγάλη μου χαρά να παρακολουθήσω τις εργασίες που οδήγησαν σήμερα στην διοργάνωση αυτή για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Είναι πολύ σημαντικό εμείς, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μεταξύ των 27 κατώμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Η αξιοσέβαστοι συνάδελφοι και βεβαίως οι θεσμικοί συνάδελφοι, μάλλον οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, είναι σημαντικό να δώσουν εδώ τη συνεισφορά του. Να μιλήσουμε για τα φαινόμενα βία που βασανίζουν αυτή τη στιγμή τι γυναίκε οι αριθμοί είναι τέτοιοι που απαιτούν να αναλυφθεί άμεση δράση για τις γυναίκες που είναι θύματα βίας ψυχολογικής και σωματικής ε, εντός και εκτός των χωρών μας. Στην Ευρώπη, στην πολιτισμένη Ευρώπη, ένα τέταρτο των γυναικών υποφέρει από ψυχολογική ε, βία τουλάχιστον, 10% και πάνω, επίσης είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Για να μην μιλήσουμε για τους αριθμούς των αυξανόμενων περιπτώσεων, και άλλων φαινομένων βίας που πλήττουν ιδίω τα κορίτσια. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και το έργο της δικής μας Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο αριθμός των γυναικών που είναι θύματα βίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που θα πρέπει να εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ακόμη να διαβεί ένα δρόμο μακρύτατο και πολύ τραχή. Το να εξαλείψουμε τέτοια φαινόμενα βίας κατά του γυναικείου φίλου είναι δύσκολο και εδώ εμείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, τις διεθνείς συμβάσεις και τις δηλώσεις πρέπει να προστατεύσουμε το πρόσωπο των γυναικών, τα άτομα συγκεκριμένα δεν μιλάμε μόνο για διακριτική μεταχείριση των γυναικών, αλλά τη βία κατά των παιδιών επίση. Ή το δικαίωμα να μην υποφέρει κανεί από απάνθρωπη ή υποβαθμιστική συμπεριφορά. Πολλέ φορέ ε, έτσι καταργούμε το πρόσωπο τη γυναίκα. Η βία κατά των γυναικών που οδήγησαν στις ε, Αποφάσει της 26ης Νοεμβρίου για την κατάργηση των φαινομένων βίας κατά των γυναικών και την απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου της φετινής χρονιάς για την ισότητα ανδρών και γυναικών είναι αναπόσπαστα τμήματα της γενικότερης απόφασης που πρέπει να λάβουμε και είναι αποφάσεις που στηρίχθηκαν από συναδέλφους όλων των πολιτικών παρατάξεων. Τον κύριο Ταραμπέλα, την κυρία Φιγκερέιδο και ούτω καθεξή. Συναδελφοί που όλοι μαζί θέλουν να καταπολεμήσουν την βία κατά των γυναικών. Ε, Κλείνοντα, Πρόεδρε, να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο συμβολικέ χειρονομίε για ιδεολογικού αγώνε, αλλά πρέπει να αναλάβουμε πραγματικέ αληθινές πρωτοβουλίε για να καταρτήσουμε κοινωνικές, και κρατικέ πολιτικέ, ώστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Εν κατακλείδη να πω ότι ήδη έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Η κατεύθυνση είναι απλή και ευθεία, αλλά δεν πρέπει να ακολουθήσουμε καμία οδό κατηφορική. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια εγκάρσια προσέγγιση για τα 4,5 χρόνια θεκτής που μας απομένουν. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής. προέρχεται από την Σουηδική Βουλή. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όταν να πω στη συνέχεια των όσων ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βία των γενικών με πρόληψη. Πριν από τρία χρόνια στη Βουλή είχαμε ένα πρόγραμμα δράση. Ε, είχε 56 διαφορετικά σημεία για να σταματήσει η βία ε, όποιος ε, ενδιαφέρεται ε, μπορώ να του δώσω ένα αντίγραφο που έχω φέρει μαζί μου. Φυσικά και ο ρόλος του κράτου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ατιμορρησία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ότι πολλές φορές υπάρχει ατιμορρησία. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις που να οδηγούν σε πιο βαριές ποινές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς το ε, δικαστικό μας σύστημα θα είναι πιο αποτελεσματικό. Η εισαγγελική δράση, η αστυνομία, η Σουηδική αστυνομία έχει ένα σχετικό πρόγραμμα ε, το οποίο απέδωσε γιατί είχαμε πολύ περισσότερες καταγγελίες. Επομένως, ε, μπορεί να υιοθετηθεί ένα σύνθημα σαν το δικό μας, το σλόγγαν ότι ε, δες το κατάγγειλέ Τώρα όσον αφορά τις ε, ποινές στέρης ελευθερίας και εδώ έχει γίνει κάποια καμπάνια ε, στη χώρα μας, οπότε γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος ε, του κράτους. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, ο επόμενος τώρα η κυρία Μποσκουρτ, ε, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη μετά από αυτά που άκουσα την Κύριε Επίτροπο, πρέπει να προσφέρουμε περισσότερη προστασία και να εναρμονίσουμε ε, το, τους ποινικού ε, κώδικες, την ποινική νομολογία. Η οργάνωση των σωμαλών γυναικών έχει γράψει γράμμα στο Υπουργείο μας αλλά και η Διεθνής Αμνηστία για να σταματήσει το φαινόμενο της, ε, του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Ε, πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε μία ενιαία προσέγγιση ενίσχυσης της προστασίας των γυναικών και της δημιουργίας περισσότερων ασφαλών σπιτιών safe houses, δηλαδή ε, ε, ενός περιβάλλοντος προστασίας όπου μπορούν να καταφύγουν οι γυναίκες και ε, όσον αφορά το θέμα του ακροτοριασμού των γεννητικών οργάνων αυτό μπορεί να καλυφθεί από, την, από το πλαίσιο της πολιτικής για το άσυλο γιατί πάρα πολλές από αυτές τις γυναίκες ετούν και άσυλο έρχονται στις χώρες μας. Θα ήθελα να μάθω πώς, ε, τι κάνουν, τι πολιτική ακολουθούν άλλες ε, χώρες. Μπορούμε να μάθουμε και πολλά από την Τουρκία που είναι μια χώρα που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης. Ευχαριστώ κύριε Μπόσκοτ. Η κυρία Μητρέα από την ε, Γερουσία της Ρουμανίας. Το σύστημα, το σύστημα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών που προσπαθεί να καταπολεμήσει τη βία κατά των γενικών δεν είναι ικανοποιητικά ανεπτυγμένο. Και πολλές φορές την πρωτοβουλία βεβαίως την παίρνουν οργανώσεις πολιτών μαζί με την ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης ε, έχουμε ένα έλλειμμα κοινωνικών υπηρεσιών ε, το οποίο μπορεί να αναλάβει την ε, συνεργασία ε, με τους αδικοπραγούντες για την αναμόρφωσή τους. Εκεί στο δημόσιο τομέα πάσχουμε. Έχουμε δυστυχώς πολλά περιστατικά και υψηλά στατιστικά στοιχεία για την οικιακή βία. Βεβαίως υπάρχει ένα σύστημα, ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας, αλλά τώρα η οικιακή βία έχει γίνει ένα πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Αυτό το διαπιστώνουμε από τις ε, υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων όπως επίσης από τις ε, καταγγελίες διατάραξης της ε, Ησυχία, ε, την ε, διατάραξη της ε, δημόσιας ασφάλειας. Μέσω αυτών των καταγγελιών διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα ε, σήματα που είναι γυναίκες ε, τελικά κατηγορούν τον εαυτό τους κρίνουν οι ίδιες ότι είναι ένοχες, ότι εκείνες φταίνε δεδομένου ότι οι αδικοπραγούντες είναι συνήθως μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον πρέπει λοιπόν να τις απαλλάξουμε από το φόβο από αυτές τις, τα αισθήματα ενοχής οι γυναίκες, επίσης πάρα πολλές γυναίκες δέχονται τη βία αυτή για να μπορέσουν να κρατήσουν την οικογένεια και τα παιδιά τους και λένε ότι το κάνω για τα παιδιά μου, ανέχομαι αυτό το φαινόμενο. Ενώ είναι λάθος, απολύτως λάθος αυτή η προσέγγιση, διότι μην ξεχνάμε ότι η βία μέσα στο σπίτι επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά τα παιδιά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η βία από πλευράς ε, συντρόφου, γιατί οι άντρες ή ε, ε, όσοι διαπράττουν το δίκημα είναι τόσο υπάρχει τέτοιος θυμός, τέτοια αγριότητα η κατανόηση των αιτιών είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολη η αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως σας είπα υπάρχουν πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών αλλά και από πλευράς κυβέρνησης έχουν υιοθετηθεί στρατηγικές. Επίσης έχουμε οργανώσει ένα δίκτυο προστασίας των θυμάτων μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών. Μα ενδιαφέρει βεβαίως η εμπειρία και των άλλων χωρών σε αυτό το θέμα. δεδομένου ότι υπάρχει 10% ε, εκπροσώπηση γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς στη Ρουμανία το 52% του πληθυσμού μας είναι γυναίκες δείχνει τι μεγάλη ανισότητα υπάρχει στην εκπροσώπηση των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η εκπροσώπηση, να ακουστεί η φωνή των γυναικών και να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Το πλαίσιο δηλαδή μέσω του οποίου οι γυναίκες έχουν δυνατότερη φωνή και ισχυρότερα δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης κρατη... μέσα στο σχολείο να ενημερώσουμε ε, τα, τα παιδιά για το φαινόμενο αυτό το οποίο πρέπει να καταπολεμηθεί και να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ισότητα των δύο φίλων και η αντιμετώπιση της βίας κατά της γυναίκας είναι θέματα ε, τα οποία συνδέονται και άρα έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόοδο. θα πρέπει να δούμε λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το οποίο συμβαίνει στο σπίτι και η διαπίστωση αυτή είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και αυτό και πρέπει να δείχνουμε σε κάποιες πρωτοβουλίες τόσο ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτό το, το, το, το κοινωνικό στίγμα. πάρα πολύ ε, εύστοχη ιδέα ήταν το να οργανωθεί η σημερινή εκδήλωση. Γυναίκες και άντρες έχουμε ευθύνη για το πρόβλημα αυτό και δεν θα πρέπει ε, να χάνεται ούτε λεπτό κάθε μέρα ε, κάποια ζωή τσαλακώνεται ε, και γι' αυτό και συγχαρητήρια την περασμένη εβδομάδα ε, στο Συμβούλιο που ενέκρινε το να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την βία μεταξύ των δύο φύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες τόσο ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση για μια τέτοια στρατηγική. Και επίσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών για τις καλύτερε πρακτικές και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ε, αυτή την κοινωνική πληγή. Συμβούλιο και Επιτροπή στο πλευρό του Ευρωπαϊκού για αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε τις χιλιάδες αυτών των γυναικών οι οποίες ε, έχουν πληγεί από το φαινόμενο της βίας. Σήμερα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να συνεχιστεί αυτό το σημαντικό έργο που έχουμε αναλάβει. Όμως η ευρωπαϊκή στρατηγική χρειάζεται, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, ε, δεν θα πρέπει να είναι μια ιδέα που έμεινε στο χαρτί, θα πρέπει να υλοποιηθεί, να γίνει πραγματικότητα και το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, θα πρέπει να κάνει κάτι και αυτό απασχολεί του περισσότερου βουλευτέ που του ε, ενδιαφέρει η υλοποίηση τη ιδέα. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Καρδιά πέρα. Ο επόμενο ομιλητή. προέρχεται από την Ιταλική Γερουσία. Κύριε Διαμαντάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς να σας ευχαριστήσω για αυτή την σημαντική συζήτηση που διοργανώσατε. Να τονίσω ότι στη χώρα μας έχουν γίνει πολλά πρόσφατα με σοβαρή εμπλοκή της δημόσιας, της κοινή γνώμης για το θέμα αυτό, καθώς και το Κοινοβουλίο και της Γερουσίας μας που κατάφεραν την έγκριση για, την, ε, για τον νόμο κατά της παρενόχλησης και με σημαντική κινητοποίηση του τομέα της δικαιοσύνης. Με ευκαιρία του G8 της περασμένης χρονιάς, μια από τις προτεραιότητες της σημερινής διάταξης που συμπεριλήφθησαν ήταν η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ήθελα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να θυμίσω ότι υπάρχουν πραγματικά, πραγματικοί αριθμοί στοιχεία που προέρχονται από το παρατηρητήριο για τα φαινόμενα αυτά που αφορούν τόσο τη διακίνηση όσο και τα σχετικά φαινόμενα της βίας. Και τελευταία διαφημιστική εκστρατεία που ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου και με αυτήν την ευκαιρία ε, αφορά δύο εφημερίδες, την Ουνιτά και μια εφημερίδα από την δεξιά παράταξη, που έχουν διευθύντριες γυναίκες τους, γυναίκες μάλλον, ε, που θα μιλήσουν ε, για φαινόμενα δίας και θα δείξουν εικόνες γυναικών που αντιμετωπίζουν και πώ μπορούν να δώσουν γλώσσε στη βία. Δηλαδή θα δώσουν συμβουλέ του τύπου αν ο σύντροφό σα ασκεί βία εναντίον σα, τον παρατήστε τον. Φύγετε. Έτσι λοιπόν πρέπει να οργανώσουμε κοινέ δράσει τόσο για να ενισχύσουμε τι γυναίκε, να τι ενθαρρύνουμε, αλλά και στην πολιτική, στον πολιτικό βίο, τον οικογενειακό, τον επαγγελματικό, τον οικονομικό, να λάβουμε μέτρα και να υπάρξουν πραγματικέ δράσει. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν μπορούν πραγματικά σε στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο να πραγματοποιήσουν εδώ ένα σημαντικό μέρο του έργου μα. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Λούνασεκ του Ευρωκοινοβουλίου. Um, Ευχαριστώ. Uh, Θέλω να απευθυνθώ στην Υπουργό Ισότητα. Προέρχομαι από την Αυστρία, αλλά εδώ και 30 χρόνια ξεκίνησε την προσπάθεια για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της βίας. Στο Τυρόλο είχαμε μια ομάδα γυναικών φεμινιστριών και σε αυτή την συντηρητική περιφέρεια της χώρας μας φτιάξαμε αυτό το καταφύγιο της γυναίκες και ευχαριστούμε την Προεδρία μια που έκανε αυτές τις, ε, ανέλαφε πρωτοβουλίε και ελπίζουμε να πάμε καλά. Έχω τρεις ε, ερωτήσεις και μία αφορά την ε, Ισπανική Προεδρία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε για ένα νούμερο το οποίο να είναι κοινό και να είναι δωρεάν, κάτι σαν το 116. και αυτό να είναι για τις γυναίκες που να είναι θύματα δουλεμπορίου, εκμετάλλευση σεξουαλική. Κάποιο ο οποίο έχει μια υποψία μπορεί να πάρει τηλέφωνο να καταγγείλει. Γιατί και, με αυτό ασχολούμαι. Για πετε μα, αξίζει τον κόπο να περιλάβουμε και αυτή την περίπτωση. Έχω τώρα άλλε δύο ερωτήσει. Πρώτα-πρώτα έχουμε μια ομάδα γυναικών, κυρία Ρέντινγκ. Μια ομάδα γυναικών που ζει με κάτω από το φόβο είναι οι λεσβείες γιατί και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι πηγή ε, βίας σωματικής ή ψυχολογικής και στη δουλειά αλλά και στην οικογένεια. Η Ισπανική Προεδρία ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια πρόταση ούτως ώστε να βοηθήσει τις ε, ε και να μπορεί κανείς να ζήσει ε, ειρηνικά ανεξάρτητα από σεξουαλική, σεξουαλικό προσανατολισμό. Τώρα κάτι άλλο. Αυτά τα οποία η γλώσσα μας αντικατοπτρίζει την κυριαρχία των ε, ανδρών. Άρα θα πρέπει να αναλυθεί μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και θα πρέπει αυτά τα οποία λέμε, οι γλώσσες, να αντικατοπτρίζουν το 50% του πληθυσμού, δηλαδή τις γυναίκες. Κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους σας. Ευχαριστώ. Ε, η επόμενη μιλήτα είναι από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, η κυρία Βίντο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Αγαπητή αγαπητά μέλη και συνάδελφοι. Εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή για τις Οικογένειες του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε αυτό το επίκαιρο θέμα. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Καταρχάς, Πόσες φορές συζητούμε αυτό το θέμα στην, ε, δημοσίως, στην κοινή γνώμη και δεύτερον, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Εμείς το νομικό πλαίσιο το ξέρουμε, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι στην καθημερινή ζωή ο κάθε πολίτης μας ε, είναι ενημερωμένος για το, τις νομικές δυνατότητες και το πλαίσιο που υπάρχει θα πρέπει και επίσης ε, δεν νομίζω ότι ακούγεται ε, καθημερινά αυτό το πρόβλημα ενώ θα έπρεπε κάθε μέρα να προβάλλεται κάθε μέρα να υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκες να δουν ότι ακούγεται η φωνή τους και ότι μπορούν να ξεπεράσουν το φόβο τους να, να καταγγείλουν, να δηλώσουν και να καταλάβουν ότι η βία εναντίον τους είναι ποινικό αδίκημα. Τα οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν το ποινικό πλαίσιο ε, και τις, ε, την, τις ποινές που προβλέπονται ε, ώστε οι γυναίκες να ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες θα ήθελα μία εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία να περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο, τον ποινικό κώδικα, ε, τις ε, παραγράφους του ποινικού κώδικα που αναφέρονται σε αυτό το θέμα και τις ποινές που επιβάλλονται. Θα ήθελα να έχω μία γενική επισκόπηση ε, όλων αυτών των στοιχείων. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, πιστεύω ότι τα ερωτήματα αυτά προς την Υπουργό Ισότητος ε, έχουν ολοκληρωθεί, ότι έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών παρόλο που όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν θα μπορέσουν να μιλήσουν στο δεύτερο γύρο. Και γι' αυτό θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό καταρχάς και να ε, ολοκληρώσω εδώ τους ομιλητές στον πρώτο γύρο θα λάβετε το λόγο. Όσοι μείνατε εκτός, ε, στο, επόμενο πάνελ θα σας δώσω το λόγο. Δίνω λοιπόν και πάλι το λόγο στην κυρία Υπουργό, στην κυρία Ίντο Αλμάγκρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα όσα είπατε και όλους όσους έλαβαν το λόγο γιατί έτσι μπορούμε τώρα να σας εξηγήσουμε πώς έχει η κατάσταση σε κάθε μια χώρα και επίση έτσι θα μπορέσουμε να αντιπαραβάλλουμε τις πρακτικές και τις εμπειρίες μας και πώς η μία μπορεί να βοηθήσει την άλλη. Οπότε, να πω κάποιες σκέψεις μου για τις ερωτήσεις που υπευλήθησαν. Αυξάνεται σε κάποιες χώρες η βία των δύο φύλων και αυτό ε, ελέγχθη από κάποιους πραγματολόγο και από την άλλη μεριά ε, έχουμε το θέμα τη αμφισβήτησης με τον Γιώργο του Παράδοση του Ζωγαλού και γι' αυτό γίνεται αυτό. Τώρα έχουμε επίσης και αύξηση όμως των ε, ε καταγγελιών. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκε εμπιστεύονται περισσότερο τα θεσμικά όργανα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση στην κοινωνία. Και έτσι έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Θα πρέπει να γίνει μια σωστή διάγνωση, θα πρέπει να ξέρουμε τις ε, πραγματικές διαστάσεις, θα πρέπει όλος ο κόσμος να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, γιατί νομίζω στην ε, ε, Ισπανία έγινε ένα βήμα. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος προβλέπει κάποιες ποινές, κάποια μέτρα, πρόληψη, κοινωνική κοινωνικού λειτουργού που βοηθάνε. Οπότε αυτό το θέμα πρόκειται να αντιμετωπιστεί σαν ένα δημόσιο ε, θέμα. Ε, να μην είναι κάτι μεταξύ ενός ζευγαριού. Είναι θέμα της κοινωνίας. Ε, όλοι έχουμε ευθύνε. Και γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικό είναι να περάσει αυτό από τα ΜΜΕ. Και εδώ στο Κοινοβούλιο είναι σημαντικό το ότι έγινε αυτή η εκδήλωση. Να υπάρξει ενημέρωση για αυτό και άλλα συναφή θέματα στην ε, χώρα μας. Αποφασιστικά έχει προχωρήσει η πολιτική μας για να αναλαβούν και οι πολίτες τον ε, ρόλο τους και γι' αυτό από το σχολείο, από τις πιο τρυφερές να ξεκινάει η ενημέρωση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και ο περισσότερος κόσμος ξέρει τι γίνεται, ξέρει για τη βία των γυναικών και το μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης. Όταν ξεκινήσαμε την ενημέρωση ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε στην, στο, να, να υπάρχουν ψευδεστήσεις ε, ε, προόδου στον, στον κόσμο και έτσι να αποκοιμιέται ο κόσμος αντί να ε, ξυπνά. Οπότε δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι απλώς έχουμε κάποια περιστατικά από το να ακολουθεί το άλλο. Πρόκειται για φαινόμενο με αιτίε και αποτελέσματα. Πρόκειται για μια εκδήλωση του φαινομένου της ανισότητας. Είναι κάτι που ανάγεται σε πάρα πολύ ε, απότερο παρελθόν. Χρειάζεται επομένω αλλαγή νοοτροπίας. Όλοι οι πολίτες, όλα τα ΜΜΕ έχουν ευθύνη. Θα πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα στα στερεότυπα στους παραδοσιακού ρόλους, αλλαγή νοοτροπίας και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έγινε μια συγκεκριμένη ερώτηση εκ μέρου ε, μια βουλευτήνα από την Αυστρία όσον αφορά αυτό το, το, το, το, το νούμερο πρώτη ανάγκη για να μπορεί κανεί να πάρει τηλέφωνο και να καταγγείλει περίπτωση βία. Αυτό περιέχεται ω συμπέρασμα στη, στο, στο, στο καταληκτικό κείμενο του Συμβουλίου Υπουργών. Όπως και το 116, επομένω έχουμε το αντίστοιχο αυτό νούμερο. Και ρωτήθηκε το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ένα τηλέφωνο που κανένας να μπορεί να καταγγείλει το, το, το δουλεμπόριο σεξουαλική εκμετάλλευση. Βεβαίως ε, υπάρχουν ε, σεξουαλικές σκλάβες ε, ακόμα και σήμερα στον 21ο αιώνα. Ε, αυτό άλλωστε το προβλέπει και ο σχετικός ορισμός του ΟΗΕ. Γι' αυτό και χρειάζεται πρόγραμμα δράση. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό το ότι θα έχει σχέδιο οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σου το βεβαιώσει και η Επίτροπο. Τον Απρίλιο κιόλα θα κατέβει αυτή η πρόταση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα ε, σύνολο μέτρων και προτάσεων. Βεβαίω και να υπάρχει ένα τέτοιο τηλέφωνο είναι πάρα πολύ θετικό, να μπορεί να αισθάνεται η κάθε γυναίκα ότι ε, προστατεύεται και ότι αν είναι θύμα σεξουαλική βία και εκμετάλλευσης μπορεί κάτι να κάνει και να ε, αντιμετωπίσουμε έτσι τις μαφίες, αυτά τα δίκτυα εκμετάλλευσης και να έχουμε περισσότερη ευαισθητοποίηση του κόσμου, των πολιτών. Γιατί κάποιο που είναι δημοκράτης δεν μπορεί να ανέχεται συνενοχή σε τέτοιες ε, μορφές δουλειά. Γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχει σιγή και συνενοχή. Άρα, μέτρα πρώτον, για προστασία των θυμάτων. Δεύτερον, δίωξη αντιμετώπιση των δικτύων και τρίτον, ευαισθητοποίηση του κόσμου και να σταματήσει η συνενοχή ή ανοχή. Άρα χρειάζεται ένα σύνολο μέτρων και δράσεων. Και να υπάρχει επομένω ε, κάποιο ε, ε, κάποιο τηλέφωνο, κάποιο θεσμικό όργανο μπορεί να προσφύγει για να ξεφύγει από, από τέτοια δίκτυα. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο Ρέντινγκ για να μας δώσει κάποιες δικές της απαντήσεις. Well, thank you, Madam Chair, and... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ εντυπωσιάστηκα από τις λεπτομέρειες που μας δόθηκαν. Ιδιαιτέρως από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Προφανώς ήδη πολλά προβλέπονται στα εθνικά, στα επιμέρους κράτη για την προστασία των γυναικών ή για την καταπολέμηση της βίας. Αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεντρώνουμε και μελετούμε όλα τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί ώστε να διδαχθούμε από όσα έδωσαν αποτελέσματα και όσα δεν έδωσαν επιτυχημένα αποτελέσματα. Έτσι θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα των κατώμελών που είχαν επιτυχημένες πρακτικές και θα αποφύγουμε τις αποτυχίες. Ήδη έχουμε δύο μελέτες που εκπορούνται αυτή τη στιγμή. Η μία συγκεντρώνει στοιχεία νομοθεσίας από τα διάφορα κράτη-μέλη και τις δυνατότητες να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθετική πρόβλεψη. Ε, εδώ η έκθεση αυτή θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο. Και η άλλη έκθεση αφορά τι βλαβερές παραδοσιακέ πρακτικέ, όπω σα είπα, τι επιζήμιε παραδοσιακέ πρακτικέ. Πώ συσχετίζονται με τον λεγόμενο πολιτισμό, κουλτούρα, που εγώ αρνούμαι να τον αποκαλέσω έτσι, διότι εγώ το έγκλημα θεωρώ ότι είναι έγκλημα ακόμη και όταν το πρόσχημα είναι η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Η μελέτη αυτή θα δημοσιευτεί τον Απρίλιο και στις 25 Νοεμβρίου στη διάσκεψη υψηλού επίπεδου θα συγκεντρωθούμε όλοι μαζί ώστε να σκεφτούμε τα χειροπιαστά, τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να προταθούν. Στην δική μου τη σκέψη πιστεύω και όπως άκουσα από πολλούς και από εσά, πρέπει να σπάσουμε το, τη σιωπή. Το μυστικό να γίνει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης ευρωπαϊκής κλίμακας Όπω κάνουμε για την πολιτική ισότητα των φύλων. Εδώ θα είχαμε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα επιτρέψει και στα εθνικά κοινοβούλια να αναλάβουν ευθύνε και να συζητήσουν τα θέματα αυτά και σε εθνικό επίπεδο. Δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο να συζητούν εδώ στις Βρυξέλλες. Όχι, πρέπει να πάμε στα κράτη-μέλη. Εκεί πρέπει να βοηθήσουμε και πρέπει να μας βοηθήσετε κι εσείς. Επίσης, τέθηκαν ερωτήματα για το τι συμβαίνει με τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις διακρίσεις ε, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών. Ε, είναι σαφής η χάρτα. Καμία διάκριση δεν επιτρέπεται λόγω σεξουαλικής προτίμησης προσανατολισμού, θρησκευτικών επιθύσεων, πολιτιστικών και ούτω καθεξής. Όχι, η γυναίκα είναι γυναίκα και πρέπει να γίνεται σεβαστή όπως και αν επιλέγει να ζει και ό,τι και αν πιστεύει. Και για την ε, γραμμή επιγόντων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει τη δυνατότητα να λειτουργεί αριθμός ε, άμεση βοήθειας 166. Μία είναι για τα αγνοούμενα παιδιά και αυτό εξαρτάται από το πώς θα βοηθήσουν εδώ τα κάτι μελη τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν εδώ δράση. Αν δεν το κάνουν, δεν θα πετύχουμε. Και επίση, εάν κάνουμε μια τέτοια γραμμή επικοινωνία και για τη βία κατά των γυναικών, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα, θα χρειαστούμε και την εθνική ε, στήριξη, να ασκηθεί πίεση στι κυβερνήσει. Μην έρχονται όλοι εδώ στι Βρυξέλλε και μα λένε ναι, ωραία ιδέα, αλλά πρέπει να υλοποιηθεί και στην πράξη. Ωραίο είναι να υπάρχει ένα αριθμό, αλλά πρέπει να υπάρχει και υποδομή πίσω από τον αριθμό κάποιος ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις. Κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να περάσει τους ενδιαφερόμενους στην αστυνομία ή να επικοινωνήσει με τα, θύματα. Δεν αρκεί ένας αριθμός λοιπόν. Εδώ πραγματικά υπολογίζω στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και να πω, Πρόεδρε, ότι αν τέτοιο νούμερο, τέτοιος αριθμός επικόντων δημιουργηθεί, θα σας ζητήσω να οργανώσετε συνάντηση των ευρωβουλευτών με τους εθνικούς βουλευτές, να οργανώσουν συντονισμένη δράση για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Και εγώ θα τη στηρίξω την όλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ενελεχείς πληροφορίες που μας δώσατε και μετά την προπαρασκευαστική μας εργασία θα επανέλθω και ελπίζω ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνάντηση ξανά στις 25 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στον πρώτο γύρο της ε, συζήτησης σήμερα. Και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Υπουργό Ισότητας για θέματα ισότητας της Ισπανίας, την κυρία Ιντο και την κυρία Ρέντινγκ, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρώτο πάνελ τη συζήτησή μα να σας θυμίσω ότι τώρα θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο, ένα δεύτερο πάνελ με την δυνατότητα όλοι οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν και πάλι το έντυπο για τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή μας για να μοιραστούμε εμπειρίες από τα διάφορα κράτη-μέλη. Και θα περάσουμε ακριβώς στο δεύτερο μέρος της σημερινής συνάντησης να καλωσορίσω την πρώτη μας ομιλήτρια. Είναι μεγάλη μου χαρά να υποδέχομαι εδώ την κυρία Ινές Αλμπέρντι, την εκτελεστική διευθύντρια του ιδρύματο Ανάπτυξης για τις Γυναίκες του ΙΕ, UNIFAM. Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Αλμπέρντι. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Αποτελεί για μένα μεγάλη χαρά να μπορώ να ε, απευθύνομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα που γιορτάζουμε την ε, Διεθνή Μέρα της Γυναίκας και ταυτόχρονα τη 15η επέτειο της διακήρυξης και της πλατφόρμας ε, δράσης του Πεκίνου. Ευχαριστώ τον κύριο Γερζιμπούζερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού και την Εύα Μπρίτ Σβένσον, την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισότητα των δύο φύλων που διοργανώσαν την σημερινή εκδήλωση επίσης. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Υπουργό Ισότητας, ε, την ε, Βιβιάννα Αίδο, αλλά επίσης και την Βιβιάν Ρέντινγκ, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια επίτροπο για τα δικαιώματα των πολιτών. Σήμερα, 15 χρόνια μετά την πλατφόρμα του Πεκίνου και επίσης δέκα χρόνια μετά την διακήρυξη για την νέα χιλιετία θα πρέπει να θυμόμαστε ε, τι πρόοδες που έχουν κάνει όσον αφορά ε, τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, είναι σήμερα 18,6% οι βουλευτίνες κατά μέσο όρο στον κόσμο και έτσι γεφυρώνεται αυτό το χάσμα. Και υπάρχει μισθολογική πρόοδος, μισθολογική ισότητα στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. παρόλα αυτά όμως μας μένουν μόνο πέντε χρόνια από τον στόχο που είχαμε τάξει όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε παρόλα αυτά και ακόμα οι γυναίκες ε, υστερούν 4 προς 1 ε, όσον αφορά τις ε, βουλές του κόσμου και δύο τρίτα των εργαζομένων γενικών έχουν πάρα πολύ ευάλωτε θέσει εργασία και πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες και είναι δεκατομμύρια οι ανήλικες και οι ενήλικες γυναίκες οι οποίες υφίστανται καθημερινά συμπτώματα βία. Παρ' όλα αυτά ε, θα πρέπει να δούμε ότι ο σημερινό μας στόχος της Διεθνής Μέρας της Γυναίκας ε, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τα επιτοβεύματα γιατί έχουμε ένα σύνολο 186 χωρών που επεκύρωσαν την ΣΕΝΤΑΒ ε, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνήσεις ε, έχουν την αρμοδιότητα και υποχρέωση να αντιμετωπίσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε κάθε περίπτωση βίας κατά γυναικών και ανηλίκων γυναικών. Ε, σε ανώτατο επίπεδο του ΙΕ αυτό εγκρίθηκε. Είχαμε την καμπάνια του Γενικού Γραμματέα που λέγεται ούνεται, ούτω ώστε να μπει ένα τέλο σε αυτό το φαινόμενο. Και 10 χρόνια πέρσι από το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου τη Ασφάλεια που αφορά γυναίκε, ασφάλεια και ειρήνη. Το δε ψήφισμα 1820 αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ε, στι διεθνεί συγκρούσει και πολέμου σαν θέμα ασφάλεια διεθνέ και καλεί σε τερματισμό της ε, ατιμορρησίας. Παρ' όλα αυτά, απουσιάζουν από τα ενευτικά πλάνα οι γυναίκες ε, όμως είναι λιγότερο από 10% των αντιπροσωπιών ε, που πάνε για τις ε, διαπραγματεύσεις ενώ παρόλα αυτά τα, τα φαινόμενα σεξουαλικής βίας κατά τους πολέμους, τις συγκρούσεις ε, έχουν αυξητικές τάσεις αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ε, πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, θα πρέπει να σας ε, ευχαριστήσω γιατί τίθεται με αυτή την εκδήλωση το πρόβλημα. Να ευχαριστήσω την κυρία Σβένσον επίσης για τις ενέργειές της, τις πρωτοβουλίες της. Πέρσι, στα πλαίσια της εκστρατείας του UNIFEM, πες όχι κατά της βίας κατά των γυναικών, εσείς εδώ εγκρίνετε αυτή την διακήρυξη που θέλει να θεσπιστεί μια χρονιά μηδενικής ανοχής. Ε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με όλες τις κοινωνικές πολιτικές. Αυτή η επομένω εκστρατεία που προείπαμε έγινε μια πλατφόρμα και έτσι είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσει κανείς το τι έχει γίνει, να αξιολογήσει αυτές τις πρωτοβουλίες, ε, προσώπων, κυβερνήσεων, νέων των πολιτών κατά της βίας. Είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην ε, εκστρατεία του ΟΗΕ. Και από τότε που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, από τον Νοέμβριο πέρσι, έχουμε πάνω από 200.000 δράσεις αυτής της καμπάνιας Πεσόχη και αυτό έχει υπερκαλύψει τον αρχικό στόχο. Ε, είχαμε πει για 100.000 ε, δράσεις για την ε, μέρα της γυναίκας. Οπότε, ε, σε 190 χώρες έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα στο διαδίκτυο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εκστρατεία, κάποιες πρωτοβουλίες που να σχετίζονται με όλες τις μερίδες της κοινωνίας. Έχουμε 200 φορείς της κοινωνίας των πολιτών που σχετίστηκαν με αυτή την καμπάνια και 69 κυβερνήσεις, 30 ε, αρχηγούς ε, κρατών και πάνω από 700 ε, βουλευτές που προσυπέγραψαν τη σχετική δήλωση συμμετοχής σε πολλές περιπτώσεις είχαμε θέσπιση αναγκαίων μέτρων, ε, όπως, όπως η απόσυρση, η διαγραφή, άρση κάποιων επιφυλάξεων για το ΣΕΝΤΑΒ, ε, η προσχώρηση στο, στο πρωτόκολλο που επισυνάβεται στη ΣΕΝΤΑΒ, το οποίο είναι ε, μη υποχρεωτικό. Επίσης είχαμε κάποιους δράσεις όπως χρηματοδότηση προγραμμάτων για περισσότερη εμπλοκή της δικαιοσύνης και της ε, αστυνομίας. Χρειάζεται επομένω να γίνουν πράξη οι διακηρύξεις, οι υποσχέσεις, να έχουμε και ένα ψήφισμα για ε, ένα φορέα που θα ασχολείται με αυτό το πρόβλημα και όλα αυτά νομίζω διατυπώνονται πάρα πολύ ξεκάθαρα στο ψήφισμα του Σεπτεμβρίου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπου έχουμε ε, ένα απολογισμό, ένα, μια, μια αξιολόγηση του όλου τοπίου, το πώς έχει η κατάσταση ε, στον ΟΗΕ για την ισορρήνωση των δύο φύλων. Και έχουμε όπως λοιπόν αυτή την καινούργια υπηρεσία, το έχει αναλάβει μια νέα αναπληρώτρια γενική γραμματέας για τα προβλήματα που αφορούν το τι μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά στα πλαίσια του ΟΗΕ. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα οικονομικών πόρων, τόσο ώστε να ξεκινήσουμε κάποιες καινοτόμες δράσεις. Και έτσι, με αυτή την καινούργια υπηρεσία θα μπορούσαμε πιο συστηματικά να, να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε σε προσπάθειες των ε, χώρων μελών έτσι θα έχουμε μια συγχώνευση των τεσσάρων φορέων που υπάρχουν σήμερα, ο Σάγι Ντάου, Ινστρό και Ουνιφέμ. Και αυτή η νέα υπηρεσία, το νέο θεσμικό όργανο, θα είναι δυνατόν να κάνει αναλύσεις, θα είναι δυνατόν να δουλεύει με τρόπο προγραμματικό, να τάσει κάποια πρότυπα για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και έτσι να προστατεύεται το κάθε δικαίωμα της γυναίκας και να περνάει μέσα από κάθε πολιτική του ΟΗΕ, του συστήματός του, ε, η ισότητα. Επίσης, έτσι θα έχουμε εποπτεία, παρακολούθηση, ε, παροχή πληροφοριών όσον αφορά το σύστημα του ΟΗΕ. Και πρόκειται για κάποια πρόκληση που προϋποθέτει ε, εμπειρία και γνώση των οργανώσεων και δικτύων για τα θέματα της ισότητας. Έτσι δόθηκε αυτή η όθηση για προστασία δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητα ε, μεταξύ των δύο φύλων από τότε που είχαμε την πρώτη διάσκεψη του Μεξικού το 1975. Πρόκειται για μια εντολή ξεκάθαρη ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την επίτευξη του στόχου για να έχουμε και έναν απολογισμό με μια εποπτεία του τοπίου αλλά θα το καταφέρουμε αυτό μόνο εάν έχουμε όλους τους πόρους που απαιτούνται. Η πλατφόρμα του Πεκίνου ε, έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει στράτευση κάθε και χρησιμοποιήσει κάθε πόρο απαραίτητο και δυνατό γιατί τώρα έχουμε αυτούς τους φορείς που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας των φύλων και έτσι έγινε κάποια προσπάθεια ε, αυτά τα χρόνια παρά το ότι υπήρχε πάγια έλλειψη πόρων και άρα ε, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το πολύ πολύ μικρό κομματάκι των πόρων του ΙΕ ε, και οι ομάδες, οι φορείς των γυναικών ευθύς εξ αρχής είπανε ότι για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που έχει αυτή η καινούργια υπηρεσία χρειάζεται έναν προϋπολογισμό ενός δις δολαρίων ετησίως. Και έτσι θα προχωρήσει η δουλειά του καινούργιου φορέα. Πρόκειται επομένως για έναν πάρα πολύ σημαντικό στόχο, αλλά όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων, έτσι θα πετύχουμε κάτι και θα πρέπει να έρθει αυτή η έλλειψη των πόρων για τις προσπάθειες κατά της βίας και έχουμε ε, μια έκθεση ενός ιδρύματος του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της βίας. Πρόκειται για ένα ίδρυμα ε, το οποίο θα βρει τους απαραίτητους πόρους για τις προσπάθειες καταπολέμησης της βίας. Πρόκειται για ένα ταμείο, για ένα ίδρυμα ε, που υπάγεται στο UNIFEM στο σύστημα του ΟΗΕ και από τότε που συγκροτήθηκε αυτό το ταμείο, το ίδρυμα ήταν ε, πάρα πολύ αποφασιστική σημασία σαν μηχανισμός για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και ανηλίκων. Πέρσι αυτό το ταμείο, το ίδρυμα έφτασε σε σύνολο ε, δεσμεύσεων πληρωμών πρικοδότηση 23,6 εκατομμυρίων δολαρίων και ε, αυτό έγινε κατόπιν μιας πάρα πολύ αναλυτικής ε, αντιμετώπισης με διαφάνεια και θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι πόροι που προοικοδότησαν σήμερα αυτό το το, το Ίδρυμα είναι ένα ποσό ανώτερο από πέρσι. Και αντίστοιχα το 2008 ήταν ανώτερο το 2007. Ε, όμως όλα είναι και περισσότερα χρήματα απαιτούν. Το 2009 ή διατυπώθηκαν 1643 ε, αιτήσει που οδήγησαν σε πρικοδότηση 857 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ από την άλλη μεριά είχε προβλεφθεί πρικοδότηση μόνο 23 ε, εκατομμύριων δολαρίων και η έκθεση που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή για τις γυναίκες του ΟΗΕ ε, διατύπωνε ότι απαιτείται πρικοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για το Ίδρυμα το 2015. Είναι αυτός ένας στόχος που επίσης υιοθετήθηκε από την καμπάνια του Γενικού Γραμματέα εν του 2015. Θα πρέπει όλο το σύστημα του ΟΗΕ να συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου και γι' αυτό και η UNIFEM ε, συνεννοήθηκε με την πρωτοβουλία Κλίντον και παρουσιάστηκαν κάποιες πρωτοβουλίες δράσεις το 2009. Ε, αυτό το Ταμείο του ΟΗΕ κατά της βίας δεν είναι ο μόνος μηχανισμός ε, που έχει ο UNIFEM ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τη βία των γυναικών. Στον υπόλοιπο χρόνο που έχω θα σας πω κάποιες πρωτοβουλίες που βγήκαν από την αναθεώρηση της πλατφόρμας του Πεκίνου συν 15 τις τελευταίες 15 μέρες. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει σε παγκόσμια κλίμακα να θεωρηθεί ότι έχουμε αυτό το στόχο και θα πρέπει να υλοποιηθούν υποσχέσεις οι πολιτικές και επομένως θα πρέπει να έχουμε περισσότερους επαγγελματίε και πολιτικούς που έχουν εμπλακεί, που έχουν πρόσβαση σε κάποιες βάσεις δεδομένων για τα φαινόμενα της βίας και αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη η UNIFEM έφτιαξε το Παγκόσμιο Κέντρο Γνώσης όπου έχουμε κάποιες εμπειρίες, κάποιες γνώσεις, κάποιες, κάποια πρακτικά ζητήματα ε, από όλο τον κόσμο. Και έτσι, με πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων, ε, αποκτά κανείς τη γνώση για να μπορεί να παρέμβει, να γίνει πιο αποδοτικός, να έχει καλύτερα αποτελέσματα ε, και να πιάνουν τόπο οι επενδύσεις που γίνονται για την πολιτική αυτή. Επί τη βάση των πρωτοβουλίων που έχουν ελευθεί, των εμπειριών που υπάρχουν για τη δίεκατα γυναικών και ανηλίκων, και προέρχονται όλες αυτές οι πληροφορίες από το Διεθνές Κίνημα το Γυναικείο, από οργανώσεις κοινωνικές, ε, κυβερνητικούς φορείς ή τον ΟΗΕ τον ίδιο. Και έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμα της ε, UNIFEM για τις ασφαλείς πόλεις ε, για να έχουμε λιγότερη παρενόχληση, λιγότερη σεξουαλική βία στη, στους δημόσιους χώρους της πόλης. Ε, ξεκίνησε αυτό από την εμπειρία στην Λατινική Αμερική, ούτω ώστε οι πρωτοβουλίε αυτές να καλύψουν μια σειρά πόλεων σε όλο τον κόσμο. Πρόγραμμα το οποίο προωθεί και τη συνεργασία και κοινοτήτων, τοπικών αρχών, αναλύει τα πρακτικά μέτρα ασφάλειας, την ε, κινητικότητα και την άμυνα. Οπότε, πρέπει η UNIFEM να συνεργαστεί και με τον ιδιωτικό τομέα ούτω ώστε να υπάρχει πιο σημαντική και μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών σε επιχειρήσεις γιατί σε διευθυντικές θέσεις υπάρχουν λίγες γυναίκες και έγινε πρόσφατα μια μελέτη του McKinsey και σε παγκόσμια κλίμακα ε, έγινε έρευνα σε 2.300 υψηλά στελέχη και Εν τρίτον από αυτούς που προτίθηκαν είπαν ότι οι πολιτικές ισότητας ε, απέδωσαν ε, κέρδη. Ε, εν τρίτον είπε ότι πρόκειται να προχωρήσουν σε τέτοιες ε, κινήσεις για περισσότερη ισότητα γιατί είναι σίγουροι ότι έτσι θα πάει καλύτερα η δουλειά γιατί θα αποδώσει η επιχειρηματική δράση. Επομένως αναγνωρίζουν και οι ότι η ισότητα των δύο φύλων κάνει καλό στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις την περασμένη εβδομάδα η UNIFEM στο, στην υπηρεσία της ε, Παγκόσμιας ε, Συμφωνίας του ΟΗΕ ε, αποφάσισε να ξεκινήσει μια, μια πρωτοβουλία για μηδενική ανοχή κατά της βίας στην εργασία. Έτσι θα πρέπει να υπάρξει κάποια εκπαίδευση του προσωπικού και των υπευθύνων ασφαλείας για να μπορούν να επισημάνουν τα ε, δείγματα της ε, εκδηλώσεις βίας. Στο Πεκίνο συν 15 την περσμένη εβδομάδα ξέρετε τι είπε η κυρία Μπριτ Σβένσον ότι είναι πάρα πολύ βασικό οι πολιτικοί να εμπλακούν στην ε, προσπάθεια αναβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ως πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών θα πρέπει να παρατηρήσω ότι πετύχαμε μια αλλαγή. Η βία κατά των γυναικών είναι μια προτεραιότητα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είπε επιλέξει η κυρία Σβένσον και ακριβώς είναι αυτό ε, που θέλουμε να καταφέρουμε με την καμπάνια δινοούνεται για τον της βίας κατά των γυναικών και ελπίζω ότι του χρόνου στην ε, Διεθνή Μέρα της Γυναίκας θα μπορέσουμε να, να πούμε πώς ε, αυτές οι πολιτικές υποσχέσεις αλλά και οι δράσεις ε, πέτυχαν να κάνουμε κάποια μετά πρόοδο κατά της ε, βίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αλβέντε και τώρα δίνω το λόγο στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος Μάρτιν Καπόφσκι, ένας δημοσιογράφος ε, από τη Βουλγαρία. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Μαρτίν Καρμπόφσκι, εργάζομαι στην δημοσιογραφία για διάφορες, ε, για θέματα ερεύνης εδώ και 15 χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για την πρόσκλησή της καθώς και όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτή. Είναι αλήθεια ότι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα το κάθε κράτο μέλο ε, έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δυστυχώ όμω μοιάζουμε και στα αρνητικά φαινόμενα. Εδώ μιλάτε για τη βία. Στη χώρα μου μιλάμε για επιβίωση, ούτε καν για βία. Δεν μιλάμε για εκστρατείε ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες επίσης χώρες κάθε, μάλλον μία στις τέσσερις γυναίκες είναι θύμα βίας. Στη Βουλγαρία τα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι η κατάσταση είναι η ίδια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω στιγμή. Δεν πιστεύω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βουλγαρία οι γυναίκε που είναι θέματα τη βία ανέρχονται στου ίδιου αριθμού. Η βία στη Βουλγαρία είναι κάτι το τελείω διαφορετικό. Σήμερα θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για το τι συμβαίνει στην πράξη πράγματα πολύ δυσάρεστα και αρνητικά. Στη Βουλγαρία δυστυχώς είμαστε μέλ, μέρος των αρνητικών παραδειγμάτων στο μεγάλο ευρωπαϊκό ε, κράτος. Μιλάμε για γυναίκες που τους έχουν ρίξει στο πρόσωπο οξύ. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος πολίτης της ευημερούσας ε, γυραιάς Ευρώπης. Εδώ δεν μιλάμε για απομονωμένα περιστατικά. Μιλάμε για επιδημία πραγματική, η οποία λαμβάνει ολόνα και μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν υποφέρουν όμως μόνον οι γυναίκες, ούτε οι εκπρόσωποι των μειονοτήτων, τα μέλη των μειονοτήτων. όσοι διαφέρουν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι, μιλάμε για απλές εργαζόμενες, νοσοκόμες, ταμείες, φοιτήτριε, γιατροί. Στην Βουλγαρία είχαμε 24 τέτοιες περιπτώσεις. Γυναίκες που τους πέταξαν οξύ στο πρόσωπο τα τελευταία 10 χρόνια. Εδώ μιλάμε για ένα είδο ε, συμπεριφορά που θεωρείται φυσιολογική στην ε, Βουλγαρία. Βεβαίω μια γυναίκα επιβιώνει επιζήματα με μια τέτοια επίθεση, όμω όχι κανονικά. Εννοείται αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στο Πακιστάν ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσως να υπήρξε μία απομονωμένη περίπτωση, στη Ρουμανία άντε άλλες δύο, όμως στη Βουλγαρία είχαμε 24. Επίσης, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και σε άνδρες. Τους ρίχνουν οξύ στο πρόσωπο και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, απαράδεκτο για μια χώρα της οποίας είμαι κάτοικος. Υπήρξε μία και μόνο πραγματική καταδίκη για τον άνθρωπο που παρήγγειλε, που έδωσε την εντολή για μια τέτοια εγκληματική ενέργεια. Συνήθως υπάρχει ο ο παραγγέλων και εκείνος που διαπράττει το έγκλημα, την ενέργεια αυτή. Το κράτος μας λοιπόν είναι απίστευτο να μην υπάρχουν πιο αποτελεσματικές ποινές. Αυτά φυσικά είναι προβλήματα που μας έχουν μείνει ως κατάλοιπα του παλιού κομμουνιστικού συστήματος. Όμως σε ό,τι φορά τις γυναίκες, η βία, τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών, αυτό θεωρείται μέρος των κανονικών οικογενειακών σχέσεων. Ακόμη και όταν μιλάμε για την ρήψη οξέως στο πρόσωπο μιας γυναίκας, η κοινωνία το αντιμετωπίζει αυτό σαν ένα θέμα προσωπικό που πρέπει να μείνει μέσα στην οικογένεια. Τα νίκο μη ενδύμω. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει εδώ, αλλά σαφώς πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το κράτος. Ήδη εδώ συζητάμε για νομοσχέδιο, πρόταση νομοσχεδίου, που να κατοχυρώνει ότι δεν θα επιτρέπεται η βία, η εξάσκηση βία ω φαλιάρα στα παιδιά. Ότι ακόμα και αυτό θα θεωρείται μορφή βία. Αυτό στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όχι στη Βουλγαρία. Μην ξεχνάμε λοιπόν, τα θύματα αυτών των αποτρόπων εγκλημάτων είναι συνήθως γυναίκες. Αυτές οι φρικτές πράξεις σκοπό έχουν να καταστρέψουν την εξωτερική ομορφιά, να τις σημαδέψουν διαβίου, να τις αφήσουν ουλές για όλη τη ζωή στο πρόσωπο. Τα τελευταία τρία χρόνια και μόνο σημειώθηκαν περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι συνήθως. Ο Πρωθυπουργό μα, ο κύριος Μπουρίσοφ, υποσχέθηκε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και υποσχέθηκε να προβλέψει θα, ε, ε, δια, ε, διαβίου κάθριξη για τους ε, υπεύθυνου αυτών των εγκληματικών ενεργειών. Μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχουν πάντοτε περιοχές στην Ευρώπη όπου η βία των γυναικών αγνοείται, την αντιμετωπίζουν σαν μέρος των ε, κλασικών οικογενειακών σχέσεων στη Βουλγαρία. Αυτό είναι ο κανόνας, δεν αλλάζει τίποτε. Ο χρόνος περνάει, τα χρόνια κυλούν, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Και αυτό που μεσολαβεί μεταξύ των συζητήσεών μας και των όσων γίνονται είναι τελικά η ζωή μας. Εδώ είναι δημοσιογράφος, δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο από το να καταγγείλω κάποια φαινόμενα. Ε, μαζί μου μάλλον γνωρίζω και έχω, έχουν ήρθει μαζί μου στι Βρυξέλλε μια γυναίκα θύμα τέτοια επίθεση, ρίψη στο ξέρω στο πρόσωπο. Άλλε πέντε γυναίκε ήθελαν να ταξιδέψουν μαζί μου στι Βρυξέλλε για να μιλήσουν για τα δικαιώματά του. Ε, γυναίκε που έπεσαν θέματα τέτοιων επιθέσεων. Οι γυναίκε αυτέ ε, θα υποβληθούν σε πλαστική εγχείρηση για να αναμορφώσουν το πρόσωπό, το του και να προσπαθήσουν να ζήσουν. Ε, τώρα, για την γυναίκα που έχει έρθει μαζί μου στι Βρυξέλλε, βρίσκεται κάπου μέσα στην αίθουσα. Δεν θα σα πω ακριβώ που κάθεται. Όμω, δεν υπάρχει ούτε ένα δημοσιογράφο στη Βουλγαρία που να μην έχει αξιοποιήσει αυτό το υλικό και να μην έχει γράψει κάποιο ρεπορτάζ, κάποιο άρθρο για αυτά τα απίστευτα εγκλήματα. Τα θεσμικά όργανα, ωστόσο, δεν αντιλαμβάνουν τι ευθύνε τους. Άγνοια και ανευθυνότητα η γυναίκα αυτή δεν έχει πλέον τα μαλλιά της, έχει μόνον ένα μάτι και σχεδόν δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανείς και να δει το στήθος της. Είναι, μιλάμε για σωματική βλάβη πλέον. Δεν θέλω να, την, ε, να σας πω ακριβώς που κάθεται. Δεν θέλω να μπορούμε να να, δεν θέλω κανείς να γίνει δακτυλοδεικτούμενος και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να επικεντρωθούμε στα θύματα αλλά θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στου δράστε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν που είναι σήμερα μαζί μα σχεδόν δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι τη, διότι ο σύζυγό τη συνεχίζει να την απειλεί. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά θα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι οι προθέσει σα και ελπίζω ότι οι προθέσεις μας θα μεταφραστούν σε χειροπιαστές ε, πράξεις. Εάν όμως η Βάγια, γυναίκα που είναι σήμερα εδώ, τολμήσει να δώσει συνέντευξη για αυτό που τη συνέβη, θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα υποφέρει χειρότερα, διότι στη Βουλγαρία οι υπεύθυνοι καμιά φορά καταφέρνουν και παίρνουν εκείνη τη θέση του θύματος Αφήστε με ένα λεπτό ακόμη παρακαλώ, λέει ο μιλητής. Δημιούργησα λοιπόν ένα κατάλογο, ένα μητρό τα τελευταία χρόνια όπου καταγράφουμε ε, τις περιπτώσεις ε, άλλων ε, εγκληματικών ενεργειών. 75 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε κέντρα περίθαλψης. Το κράτος όμως δεν κάνει τίποτα για όλα αυτά. Λέγομαι Μαρτίν Καρμπόφσκι και σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ. Και δίνουμε τώρα το λόγο στον Μόρτεν Κέρουμ, ο οποίος είναι Διευθυντής του Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην διάσκεψή μας, κρόασή μας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Γυναικείων Υποθέσεων και Ισότητος για τη διοργάνωση αυτής, αυτού του πάρα πολύ, της πάρα πολύ σημαντικής ακρόασης με θέμα την βία κατά των ε, γυναικών. Έχουμε υπολογίσει ότι περίπου 45% όλων των γυναικών στην Ευρώπη κάποια στιγμή υπήρξαν θύματα ανδρικής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, έχουμε εκτιμήσει ότι το συνολικό κόστος της βίας, της οικονιακής βίας στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι αυτές οι, αυτή η κακοποίηση θα πρέπει να θεωρηθούν ως μορφές αντρικής βίας κατά των γυναικών επειδή ακριβώς είναι γυναίκες λόγω του φίλου τους. Και αυτή η ανδρική βία κατά των γυναικών εμποδίζει την εξέλιξη των γυναικών στη δημόσια και ιδιωτική ζωή. Δηλαδή η βία αυτή αποτελεί τη παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της γυναίκας, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα της αξιοπρέπειας, ε, της ακαιρεότητος ε, σωματικής και πνευματικής, το δικαίωμα της ζωής και της ισότητος. Άρα λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αντρικής βίας κατά των γυναικών ως εμπίπτων στα θεμελιώδη δικαιώματα, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τι πρόοδος έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς έχει θεωρηθεί ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα ε, στο χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος ε, είναι τώρα δεσμευτικός βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Οι ανισότητες στις αμοιβέ ε, αποτελούν ένα κεντρικό σημείο συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να προωθήσει την ισότητα αυτή όχι μόνο στις αμοιβέ, αλλά και στο δικαίωμα εργασία, στις προσλήψεις και στην παροχή υπηρεσιών όπως φροντίδα των παιδιών αυτές όλες οι υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών μπορούν να διευρύνουν τις δυνατότητες των γυναικών να διάγουν ε, μια ανεξάρτητη και δραστήρια ζωή και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Επίσης μπορούν να τις απελευθερώσουν από σχέσεις όπου υπάρχει κακοποίηση. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε και να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο της ανδρικής ε, βίας κατά των γυναικών. Είναι γεγονός ότι το θέμα αυτό της διάστασης του φύλου δεν έχει ακόμα πλήρως ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και στη, στη διάταξη, στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες βεβαίως μιας αυξημένης συνειδητοποίησης θεμάτων ρατσισμού ε, και θεμάτων διακρίσεων, θεμάτων καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως σκεφτείτε το εξή. εάν ένας εργαζόμενος που προέρχεται από μια ε, εθνότητα πληρώνεται 15 με 20% λιγότερο από έναν άλλον εργαζόμενο ο οποίος δεν προέρχεται από μια εθνοτική μειονότητα, τότε μιλάμε και αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό ταχύτητα, ταχύτατα ως ε, ρατσισμό. Υφίσταται διάκριση ρατσιστική. Όταν όμως μια γυναίκα που εργάζεται κάνει την ίδια δουλειά με έναν άντρα και πληρώνεται λιγότερο, το εξηγούμε αυτό πολύ εύκολα επειδή έχει άλλα καθήκοντα, καθότι είναι μητέρα, δουλεύει με μερική απασχόληση και ούτω καθεξής. Άλλα διάφορα επιχειρήματα. Δεν αναγνωρίζουμε τις, τα πραγματικά εμπόδια και τις πρακτικές διάκρισης κατά των γυναικών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλους τους τομείς της εργασίας. 35 χρόνια λοιπόν έχουμε ε, επιτύχει διάφορα μέτρα ενίσχυσης της ε, θέσης ε, των γυναικών και της προστασίας τους αλλά τι συγκεκριμένα έχουμε κάνει για την αντιμετώπιση της ανδρικής βίας. Κυρία Πρόεδρε, κατά τη δεκαετία του 90 η Ευρωπαϊκή Κομισιόν και το Κοινοβούλιο αναγνώρισε το συγκεκριμένο πρόβλημα της ανδρικής βίας κατά των γυναικών Κοιτώντας όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 σήμερα, βλέπουμε διάφορα σκόρπια μέτρα, διάφορα νομικά πλαίσια ε, μη συντονισμένα, τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους ε, και είναι σκόρπια και διασπαρμένα. Αυτή η κατάσταση μοιάζει με μία κληροτίδα ε, νομική. Ενώ εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εναρμονίσουμε, να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα, τις νομικές ε, διατάξεις ε, για την ενίσχυση της προστασίας των γυναικών. Όλο αυτό το διάσπαρτο πλαίσιο δείχνει ότι η βία κατά των γυναικών, η αντρική βία δεν λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη όσο τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν έχουν ε, ωφεληθεί από την, ε, από την ισότιμη προστασία οι γυναίκες έναντι των ανδρών. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε το πρόβλημα αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έχουμε το παράδειγμα του ψηφίσματος του Μαρτίου 2009 για την καταπολέμηση της κλειτοριδοεκτομής και τον Νοεμβρίου 2009 το ψήφισμα για την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνει όλες τις μορφές της βίας. Η χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ισπανική Προεδρία έχει αναλάβει ενεργό ρόλο πάνω στο θέμα αυτό και το Ίδρυμα Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημειώσει το ενδιαφέρον της Προεδρίας για την ε, προτινόμενη οδηγία ε, ευρωπαϊκής ε, προστασίας των θυμάτων βίας η οποία φύλλεται στη διάσταση του φύλου η οποία οδηγία θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να λάβουν ισχυρά και βρία μέτρα προστασίας των θυμάτων βίας. Επίσης ε, υπάρχει πρόταση δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την, ε, το θέμα της βίας το οποίο οφείλεται και βασίζεται στη, στο φύλλο, στη, διάκριση του φύλλου. Παράλληλα, η Κομισιόν έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κατάστασης των θυμάτων και συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού θα πρέπει λοιπόν η πολιτική μας να εστιάζεται πάνω στα θύματα και να μπορούμε να υιοθετούμε απαντήσεις, αντιδράσεις και λύσεις οι οποίες βασίζονται στο φύλλο, επικεντρώνονται στο φύλλο. Το πρόγραμμα της ε, χόλμης ε, έχει ε, εδραιώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπισης και προστασίας των θυμάτων. Για να μπορέσουμε όμως να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία. Στα στοιχεία τα οποία περιγράφουν το εύρος του φαινομένου. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, συλλέγουν στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει ένα συγκριτικό ε, πλαίσιο, μια συγκριτική στρατηγική ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε όλα αυτά τα συλλεξέντα στοιχεία από τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα διαρθρωτικό ε, φαινόμενο αυτό, το οποίο καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και εδώ βέβαια μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο το Ίδρυμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το Ίδρυμά μας έχει ανταποκριθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2009, το οποίο καλεί το Ίδρυμά μας να ε, συλλέξει και να εκδώσει αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές ε, που θα καλύπτουν το θέμα των διακρίσεων γενικά αλλά και συγκεκριμένα τη βία κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το Ίδρυμα Θεμελιωθών Δικαιωμάτων έχει ε, ε, ταυτοποιήσει ε, το θέμα του φίλου ως ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τα ανθρώπινα, από τα ανθρώπινα σεμελιώδη δικαιώματα και άλλα θέματα τα οποία καλύπτονται από και μελετώνται από την υπηρεσία μας, από το Ίδρυμά μας είναι η εμπορία παιδιών, μειονοτικές εθνότητες, μεταναστευτικοί πληθυσμοί, πνευματικές ασθένειες και αναπηρίες, άτομα με ειδικέ ανάγκες. Πρόσφατα ε, δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα μιας ε, μελέτης που κάλυπτε ε, μειονότητες και διακρίσεις ε, EU MIDIS ε, λέγεται αυτή η μελέτη ε, και για να την συντάξουμε μιλήσαμε, κάνουμε συνεντεύξεις με πάνω από 23.500 πολίτες από εθνικές μειονότητες και μεταναστευτικές ομάδες. Αυτό το πρόγραμμα ήταν πραγματικά ριζοσπαστικό και μας ωφέλησε πάρα πολύ διότι συλλέξαμε μια τεράστια εμπειρία με ένα, μια πληθώρα στοιχείων και, ε, και για γυναίκες βεβαίως και τις διακρίσεις που υφίστανται στην καθημερινή ζωή ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, συλλογής και ε, έκδοσης στοιχείων τα οποία αφορούν εθνοτικές μειονότητες, γυναίκες και μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Και θα εκδώσουμε την πρώτη μας μελέτη συγκεκριμένα για το θέμα της αντρικής βίας κατά των γυναικών το 2011. Γι' αυτό έχουμε ως στόχο να παρουσιάσουμε δείκτες συγκριτικών στοιχείων για όλα τα 27 κράτη-μέλη ε, στο θέμα της αντρικής βίας κατά των γυναικών. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα μελετηθούν και θα συγκριθούν βάσει των δικτών, θα προσφέρουν αυτές ε, μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης στα ευρωπαϊκά ιδρύματα, στους φορείς και στα κράτη-μέλη, τα οποία θα επιτρέψουν όλους τους ενδιαφερόμενους να υλοποιήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά μέτρα. Τώρα, ε, εξετάζοντας το παρελθόν, ε, πρέπει να πω ότι έχουμε επιτύχει, ε, έχουμε, κάνει, έχουμε λάβει ορισμένα μέτρα τα οποία ήταν επιτυχημένα για την ενίσχυση της ισότητας ανδρών γυναικών. Όμως έχουμε ακόμα πάρα πολύ μεγάλη πορεία μπροστά μας. Εμείς υποστηρίζουμε τις, περαιτέρω, την περαιτέρω μελέτη αυτού του θέματος και ιδίως όλα τα θέματα που αφορούν τη διάσταση του φύλου, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών γυναικών και την παροχή προστασία σε περίπτωση ε, όπου είναι θύματα αντρική βία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά τους τρεις ομιλητές μας του δεύτερου πάνελ και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. και να σας θυμίσω, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε να εγγραφείτε στον κατάλογο των μιλητών απλώς συμπληρώστε το έντυπο που έχετε στο έδρανό σας και θα προσθέσουμε το όνομά σας στον κατάλογο των μιλητών. Το πρώτο... Η πρώτη μιλήτρια θα είναι η κυρία Σίνκλερ το πρώτο μέλος του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. κυρία Σίνκλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κάθε ευκαιρία συζήτηση αυτού του θέματος σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιοδήποτε φορέα είναι εξαιρετικά σημαντική. Συγκινήθηκα πραγματικά από τα σχόλια του κυρίου Καμπόφθη και από αυτά τα οποία ελέγχθησαν σήμερα εδώ. Η μάχη κατά ε, της βίας ε, που προέρχεται από άντρες είναι μία μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Σήμερα κάνω μία έκκληση στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο Ενωμένο Βασίλειο να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή καταγραφής των επεισοδίων αυτών ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο και επίσης να λάβουν μέτρα ενθάρρυνσης των θυμάτων να καταγγείλουν τα συμβάντα. Επίσης ζητώ από τα ε, κράτη-μέλη να οργανώσουν μια εκστρατεία με στόχο τη νέα γενιά, τους νέους, για να τους ενημερώσουν σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα συμφωνούμε ότι η βία είναι εντελώς απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ ήμουν σήμα βία στις 12 Ιανουαρίου 2005, έξι άντρες με γροθοκόπησαν, με ρίξαν στο έδαφος, με κλωτσούσαν και όταν πήγα βεβαίως στο νοσοκομείο είχα 21 μόλοπες και, και, και, και διάφορες, διάφορα άλλα βεβαίως προβλήματα στην υγεία μου και πού έγινε αυτό έγινε στο χώρο εργασίας μου και ποιος ήταν ο χώρος εργασίας μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα κατά αυτού του συμβάντο που έγινε εναντίον μου και ακόμα συναντώ του ανθρώπους αυτού, οι οποίοι με γρονθοκόπησαν και ε, με, ενοχλεί, με, ενοχλεί αφάνταστα αυτό, αυτό το θέμα. Ε, και με τραυματίζει βεβαίως. Ευχαριστώ κυρία Σίγκλερ. το, το, η, κυρία είναι εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με μεγάλη μου χαρά σήμερα να απευθυνθώ σε όλους εσάς μέρος της ε, συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι, με έναν δρόμο ελπίδες για όλες αυτές τις γυναίκες που υφίστανται την ιδέα μεταξύ των δύο φίλων. Εμείς ε, Είμαστε αποφασισμένοι από κοινού να αναλάβουμε δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, Συμβούλιο τη Ευρώπη, ούτω ώστε να καταγγείλουμε και καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη, εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την καταπολέμηση κατά της βίας κατά των γυναικών. Σήμερα δε το Συμβούλιο τη Ευρώπη ε, ε, επεξεργάζεται ένα κείμενο το οποίο αφορά το ίδιο πρόβλημα και πιο συγκεκριμένα την βία στο σπίτι, στην οικογένεια, για να μπορέσει να καλύψει τι γυναίκε αυτέ που πέφτουν θύματα αυτή τη βία. Θα ολοκληρωθεί αυτή μα η προσπάθεια ε, τέλος τη άνοιξη του 2011. Οι άξονες που κινούμε θα είναι πρώτον προστασία, ε, τιμωρία, πρόληψη και πώ θα ενταχθεί σε όλες τις ε, πολιτικές ισότητα και γυναικών. Και η κοινοβουλευτική μα συνέλευση ζητεί δέσμευση τη Ευρώπη να μπει ψηλά ο πύχης. Συγκεκριμένες πολιτικές. Να τοποθετηθούμε όλοι, όπως η συνέλευσή μας, και εδώ μπαίνει ο ρόλος των 47 Εθνικών Κοινοβουλίων και της κοινοβουλευτικής μας συνέλευσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν νόμους, να κάνουν στατιστικές μελέτες και να προβληθεί περισσότερο το πρόβλημα της βίας και έτσι η σχετική ε, σύμβαση να προσυπογραφεί από όλους. Από πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια και στην ε, Υπουργό Ισότητας που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχαρητήρια γιατί έτσι κάνατε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της βίας. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σε σχέση με τη συνέχεια των προτάσεών σας ε, υπό το φως της νέας συνθήκης της Λισαβόνας. Συνάδελφοι βουλευτές, θα πρέπει με μία φωνή να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Οι γυναίκες χρειάζονται να είμαστε εμείς αποφασιστικοί, να κάνουμε ό,τι πρέπει για να θεσπιστούν νόμοι και να αλλάξουν οτροπίες να έχουμε κοινό αγώνα και να έχουμε φιλόδοξους στόχους για την κατολύνση αυτής της βίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα στο χώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε χρειάζεται να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και η κοινοβουλευτική μας συνάλευση, κατά κλείδι πρόεδρε, πρέπει να σα πω ότι είναι αποφασισμένη να συνεχιστεί ο διάλογο και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε μαζί να βάλουμε ένα φραγμό στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Είναι καθήκον αυτό για όλους. Θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα για τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Ε, και εμεί προσδοκούμε να συνεχιστεί η συνεργασία με την κυριολεκτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ο επόμενο ομιλητή τώρα. Η κυρία Τόμσον, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Βουλίου. Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας για την ε, γραμμή, ε, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 116 ε, και την ιδέα για το το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σε μια ειδική ομάδα γυναικών που είναι θύματα βίας. Εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από μερικά χρόνια Στήσαμε μία έκθεση για την κατάσταση των ε, γυναικών μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες και είπαμε ότι η πιο ευάλωτη ομάδα ε, μεταξύ όλων των γυναικείων ομάδων είναι οι γυναίκες ε, μετανάστριες ε, και το Ισπανικό Υπουργείο έχει εκδώσει μια συναφή μελέτη που καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες γυναίκες μετανάστριες είναι θύματα βίας από γυναίκες με την ηθαγένεια της χώρας υποδοχής. Έχουμε ακούσει και από άλλες χώρες για τις διάφορες ομάδες το Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη όπου η έκθεση στη βία ορισμένων γυναικείων ομάδων είναι περισσότερη από τις άλλες. Ε, επίσης έχουμε ακούσει για το φαινόμενο των, ε, των ταχυδρομικών αποστολών ε, γυναικών ως νύφες προς παντριά δηλαδή, κατά παραγγελία, που οι γυναίκες αυτές παντρεύονται όχι. δικούς ανθρώπους από τη χώρα τους, αλλά παντρεύονται άντρες, ας πούμε, από την, ε, το, το ή ακόμα και στη Δανία. Είναι γυναίκες από τρίτες χώρες, ε, οι οποίες επιλέγονται μέσω όπως λέμε, ας πούμε, ταχυδρομείου, διαδικτύου, έρχονται στις χώρες αυτές λοιπόν και δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν φωνή, υφίστανται διακρίσεις και πολλές φορές θύματα βία, είναι σήματα βίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία για τη βία κατά των γυναικών έτσι ώστε να προσφέρουμε την απαραίτητη προστασία σε αυτές τις γυναίκες αλλά και για να επιβάλλουμε κοινά πρότυπα στην Ευρώπη για την προστασία των γυναικών και κοινά πρότυπα για την τιμωρία ε, των ε, δικαιοπραγούντων. Γιατί και εγώ βεβαίως εντυπωσιάστηκα, ταράχτηκα με αυτά που, που, μας είπε ο Βούλγαρος ε, ε, ο καλεσμένος μας και ρωτώ γιατί ο άντρας, η σύζυγη αυτών των γυναικών, η σύντροφοι δεν είναι στη φυλακή. Ευχαριστώ κυρία Τόμψον. Ο επόμενος ομιλητής είναι... Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Αντιπρόεδρος Μόρις Σέτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε τη σημερινή συζήτηση. Θα πρέπει να ακούσουμε και για συγκεκριμένες αληθινές περιπτώσεις Πράγματα που συνέβησαν στην πραγματικότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μένουμε κοντά στην πραγματικότητα. Και στα πλαίσια της καταπολέμησης της βίας βλέπουμε ότι πρέπει να περάσουμε και από την ομοθεσία, τον συντονισμό όπως προείπατε, τις στατιστικές και το συσχετισμό των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών, την ε, πρόβλεψη ποινικών μέτρων συνεκτικών για να δείξουμε στο σύνολο του πληθυσμού ότι υπάρχει βούληση, αμετάκλητη βούληση των θεσμικών οργάνων να αναλάβουν δράση, ότι κανείς δεν μπορεί να διαφύγει από αυτήν την βούληση. Συντονισμός Κοινοβουλίου, Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρώπης απαιτείται εδώ. Όμως ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Δύο σημεία γιατί εγώ η ίδια τα έχω ζήσει στην ζωή μου στο παρελθόν. Το πρώτο πρόβλημα ε, που έχω ζήσει από κοντά και μου φαίνεται σημαντικό είναι ότι εργαζόμαστε από κοινού για να επιτρέψουμε στις γυναίκες να υψώσουν τη φωνή τους. Οι γυναίκες που είναι θύματα βίας είναι γυναίκες που συχνά αισθάνονται ενοχές, έχουν μεγάλη δυσκολία να αρθρώσουν το τι έχουν ζήσει. Φοβούνται φοβούνται ότι θα τις ε, δείχνουν στη συνέχεια με το δάχτυλο ότι θα τις ξεχωρίζουν στο κοινωνικό τους περίγυρο. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα, τα πιο καυτά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί. Διότι όσο και να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία, οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να μιλούν, να, την, να δίνουν ε, και ένα λεκτικό περιεχόμενο στη βία που έχουν ζήσει. Είναι λοιπόν σημαντικό εδώ αυτό το μείζον πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα ένας, μια γραμμή επικοινωνίας να βοηθήσει, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Εδώ το έργο που μας απομένει λοιπόν είναι νομίζω δύσκολο. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πρώτα οι γυναίκες να πέφτουν θύματα βίας για να αντιλαμβανόμαστε στη συνέχεια τι μπορεί να είναι βία. Πρέπει να ενημερώνονται οι νέοι και οι νέες όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Κάποιος μίλησε για νεαρές κοπέλες. Εγώ μιλάω για παιδιά, διότι στον επαγγελματικό μου βίο είδα παιδιά 11 χρονών που μετά από συζήτηση ή ενημέρωση συνειδητοποιούν ότι τις έχουν πέσει θύματα βιασμού και από διετία ή τριετία. Πρέπει τα παιδιά λοιπόν αυτά πολύ νωρίς να πληροφορούνται τι είναι η βία. Να αντιλαμβάνονται τι είναι το φυσιολογικό και τι είναι παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Διότι όσοι διαπράττουν τις εγκληματικές ενέργειες νομίζουν ότι και παριστάνουν ότι διαπράττοντας βία, τέτοια φαινόμενα βίας, ασκώντας βία, παραμένουν μέσα στο κανονικό πρότυπο. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά από νωρίς από το σχολείο να μαθαίνουν την βία, ώστε να μπορούν να την καταγγείλουν. Επιμένω εδώ, διότι μου φαίνεται ότι είναι ένα σημείο σημαντικότατο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε διαρκώς οι γυναίκες να πούν κάτι. Πρέπει να εκριζώσουμε το πρόβλημα εκεί που ξεκινάει. Να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του δηλαδή. Και θέλω όλοι να συνειδητοποιήσουμε μαζί ένα πράγμα. Εργαζόμαστε σκληρά και στο Κοινοβούλιο και υπό τη δική σας την Προεδρία, κυρία Στίβενσον, εργαστήκαμε. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των γυναικών η πρόοδος στην ε, βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία δεν είναι ένα πρόβλημα που προέκυψε χθες. Σε διάφορες ιστορικές περιόδους οι γυναίκες τύχαναν σεβασμού, ήταν ε, μέλη αξιοσέβαστα της κοινωνίας. Και υπήρχαν και περίοδοι ε, που αυτή η θέση υπονομευόταν. Τίποτε δεν είναι κεκτημένο πέραν των παρατηρητηρίων που μπορεί να ιδρύσουμε. Πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση διαρκής, σταθερή, μόνιμη. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Σαρκέ. Νομίζω ότι το συμπέρασμά σα ήταν πολύ καλό. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Και επίση ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγή. Πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το έχουμε πάντοτε αυτό κατά νου. Μπορούμε να αλλάξουμε την ε, κατάσταση ως έχει. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γκουρμάη, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους ε, τους ε, παρόντες και ιδίως ε, τους συναδέλφους από την Ουγγαρία, τους συναδέλφους μου. Έχω και μία ομάδα προσκαλέσει εδώ, 25 άτομα από την Ουγγαρία, επί τη ευκαιρία αυτής της επαιτειακής ακρόασης και τους καλωσορίζω. Είναι βεβαίω αυτονόητο ότι η Επιτροπή μας έχει μία πρόεδρο με προοδευτικές ιδέες και πολύ δυναμική, διότι εμείς θέλουμε να προβάλλουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πολλές φορές κρύβεται, είναι σιωπηλό, δεν ακούγεται και θέλουμε να το βγάλουμε από αυτή την κρυψώνα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ταπατέρο, έχει πει, δήλωσε σε αυτό το κοινοβούλιο ότι η Ισπανική Προεδρία θα έχει ως θέμα προτεραιότητα την ισότητα ευκαιριών ανδρών γυναικών και την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την κυρία Αλμπέρτη, Αλμπέρτη ε, πριν από δύο εβδομάδες ε, είχαμε λάβει μέρος σε αυτό το φόρουμ, σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Συνεχώς προβάλλεται το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά. Έχω πια βαρεθεί να ακούω αυτή τη δικαιολογία. Ε, πρέπει να τα βρούμε Όπου δεν υπάρχουν πρέπει να τα βρούμε. Γι' αυτό και η έκθεση της ε, ε, UNIFEM αλλά και όλες οι εργασίες είναι πολύ σημαντική αλλά και οι εργασίες της συναδέλφους μου κυρίας Ρουίντο. Ελπίζω να παρουσιαστεί το σχέδιο οδηγίας το οποίο Μα έχει υποσχεθεί η Ισπανική Προεδρία. Βεβαίω χρειάζομαι και αυτό τον αριθμό πρώτων βοηθειών, τον 116, ε, και ε, τον, ε, είναι βεβαίω ένα αριθμό πρώτη βοήθεια που μπορούν να καλέσουν τα θύματα για την προστασία του και για καταγγελίε. Είναι πεποίθησή μου ότι όλα αυτά τα θέματα και αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετικά σημαντική η βία κατά των γυναικών είναι γεγονός στην πραγματικότητα και γι' αυτό είναι σημαντικό ότι δεν είναι μόνο γυναίκες παρόντες σε αυτή την αίθουσα, είναι και άντρες. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι χρειαζόμαστε τους άντρες στην, στον αγώνα αυτό ως συνεργάτες, ως εταίρους, ισότιμους εταίρους. Υπερβολικός αριθμός γυναικών είναι σήματα οικιακής ε, βίας, οικονιακής βίας και δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι τραγικές επιπτώσεις, οι ζημιές ε, που διαπιστώνονται από αυτήν την ε, κατάσταση. Και επίσης λέω πώς είναι δυνατόν ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει θύμα τέτοιας άγριας βίας όπως ακούσαμε από τη συνάδελφό μας ε, το να γράφουμε ε, προσυστάσεις ε, δεν ωφελεί το να δημοσιεύουμε εκθέσεις δεν ωφελεί αν δεν μεταφράσουμε τα λόγια σε πράξεις από τότε που υπάρχει συνθήκη της Ρώμης μισό αιώνα ε, υποτίθεται ότι πρέπει να έχει επιβληθεί η ισότητα. Η Επιτροπή μας πρέπει να κάνει το παν, αλλά και η κυρία Ρέντινγκ, η κυρία Επίτροπος πρέπει να εξασφαλίσει ε, την προβολή αυτού του θέματος, ώστε από προσωπικό ιδιωτικό πρόβλημα να γίνει δημόσιο πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουμε τις νοοτροπίες και να μην υποτιμούμε το λόγο του ποινικού κώδικα. Πρέπει να ποινικοποιηθούν περαιτέρω οι ποινές, να υψώσουμε τις ποινές, να γίνουν πολύ πιο αυστηρές βάσει του ποινικού κώδικα. Επίσης αυτό το, τον αριθμό πρώτης βοήθειας πρέπει να το γνωρίζουν όλα τα σήματα, ε, πρέπει να δημοσιοποιηθεί ευρύτατα Ευχαριστώ λοιπόν την Ισπανική Προεδρία για τις ε, ενέργειές της και ελπίζω και η κυρία Επίτροπος να άκουσε ε, το μήνυμά μας. Χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία σε αυτή τη θητεία του σώματος. Εάν μιλάμε για το 20% των γυναικών, 25% που είναι θύματα βίας, πρέπει όλοι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συγκεράσουν τις, τις ενέργειές τους. Κύριε Γκουρμά, ευχαριστούμε, η Πρόεδρος. Ο επόμενος τώρα ο μιλητής προέρχεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κυρία Τσαούση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Η συνάδελφός μου, κυρία Κόλια, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και εγώ σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να συμμετέχουμε σε μια τόσο σημαντική συνδιάσκεψη το θέμα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών συζητήθηκε πολλές φορές στην ε, ειδική μόνιμη επιτροπή ισότητας νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου η οποία εξέδωσε τα συμπεράσματά της σε έκθεση τα οποία μπορούμε να σας καταθέσουμε για τα πρακτικά της συνδιάσκεψης. επιπλέον την προηγούμενη δευτέρα στις 8 του μάρτη πραγματοποιήθηκε μεγάλη ημερίδα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο όπου συμμετείχαν όλες οι γυναικείες οργανώσεις ε, της ελλάδας. στην ε, ελλάδα αρμόδιο για θέματα ισότητας είναι το υπουργείο δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο από τον νοέμβριο του 2009 εξήγηλε το Εθνικό Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013 το πρόγραμμα αυτό αναλύεται αφενός σε δράσεις πρόληψης του φαινομένου και υποστήριξης των θυμάτων και αφετέρου σε νομοθετικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας έχει καταρτήσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ε, περιλαμβάνει το πρόγραμμα οριζόντιες και κάθετες δράσεις. Οι κυριότεροι άξονες ε, είναι η δημιουργία μιας τηλεφωνικής γραμμής SOS, 24 ώρες λειτουργίας, η υλοποίηση ολοκληρωμένης δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνει ημερίδες ευαισθητοποίησης θεματικό συνέδριο ενημερωτικά έντυπα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ κεντρική ιστοσελίδα και μπάνερ σε ιστοσελίδες οι κάθετες δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία 12 νέων συμβουλευτικών κέντρων στις αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας και τη δημιουργία 12 ξενώνων επίσης στις αντίστοιχες περιφέρειες σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι πρώτη φορά εκπονείται στην Ελλάδα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με πλήρη χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και το πρόγραμμα αυτό θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη ω το αρμόδιο καθήλυν Υπουργείο για την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων είναι σε θέση να βελτιώσει και να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών βία κατά των γυναικών και στο πλαίσιο τη αναθεώρηση του ποινικού κώδικα θα εξεταστούν οι νόμοι για την ενδοοικογενειακή βία, ο νόμος για τον βιασμό και την εμπορία ανθρώπων, διακίνηση γυναικών, άμεση προτεραιότητα επίσης αποτελεί η επικύρωση της σύμβασης του συμβουλίου της ευρώπης για τη δράση κατά της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων του 2005. ταυτόχρονα συμμετέχουμε στην ad hoc επιτροπή του συμβουλίου της ευρώπης που επεξεργάζεται σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη όλων των μορφών βίας που παραδοσιακά υφίστανται οι γυναίκες Τελειώνοντα, θα ήθελα να σα μεταφέρω τι ευχέ του αρμόδιου Υπουργού μα, του κ. Κατσιφάρα, και να τονίσουμε την ε, διάθεσή του για πιο στενή συνεργασία. Και προσωπικά να, να σας πω ότι θα φύγω από τις Βρυξέλλες με τα πιο θετικά ε, συναισθήματα και μηνύματα ε, καθότι σαν ε, κοινωνική λειτουργός αντιμετωπίζοντας πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στα 20 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής η αποφασιστικότητα της κυρίας Επιτρόπου ε, με έκανε να νιώσω ότι αν δουλέψουμε όλες και όλοι μαζί πραγματικά θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο της βίας. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ε, η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γιουρόκα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητος. Ευχαριστώ. Ε, σας, σας ε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, διότι θα πρέπει να συζητήσω, να φύγω και να συζητήσω με τον Επίτροπο. Είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση. Γι' αυτό θα σήξω ένα μόνο θέμα το οποίο συζητήσαμε στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Ισότητος. Το οποίο είναι το εξή. Πολλαπλές διακρίσεις ε, ε, ε, σημειώνονται κατά γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας και ιδίω κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, με πληθυσμιακές ομάδες γυναικών μεγαλύτερη ηλικίας αλλά και γυναίκες με ειδικέ ανάγκες. Αυτές οι ομάδες υφίστανται περισσότερες πολλαπλέ διακρίσεις. Επίσης, δεδομένου ότι έχω εργαστεί στι κοινότητε των Ρωμά εδώ και 15 χρόνια, διαπιστώνω μία υποβάθμιση ε, ε, των πνευματικών τους ε, ικανοτήτων καταραίουν οι γυναίκες αυτές και ψυχικά Γι' αυτό όταν ψηφίσαμε, κάναμε, υιοθετήσαμε το ψήφισμα για τους Ρωμά, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην πατριαρχική δομή αυτών των οικογενειών και στην δεσπόζουσα θέση του άντρα, του πατριάρχη σε αυτές τις οικογένειες. Έτσι λοιπόν υφίστανται διακρίσεις και λόγω της φτώχειας και λόγω της πατριαρχικής κονιακής ε, δομής και λόγω της απόλυτης ανεργίας που υπάρχει εδώ και μια γενιά, ίσως και περισσότερες αυτές τις κοινότητες. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο σωματική βία αλλά και ψυχική βία την οποία αισθάνονται. Και ε, πιστεύουμε ότι η ένταση της, ε, των επιπτώσεων διπλασιάζεται λόγω αυτού του συνδυασμού σωματικής και ψυχικής βίας. Γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε ε, τη βοήθειά σας για να μας ενισχύσετε στο θέμα των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε αυτές τις εθνοτικές μειονότητες και σε αυτές τις ε, πολύ περιθωριακές ομάδες. Μάλιστα, πολλές φορές ε, οι ομάδες αυτές κατηγορούνται ότι είναι βίες κοινωνίες, βίες ε, πληθυσμιακές ε, μειονότητες, παραδείγματο χάρη η Ρωμά, ο πληθυσμός των Ρωμά. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Στην Ουγγαρία ένα τρίτο του πληθυσμού ζει υπό φτώχε φτώχες και το 1 τρίτο του 1 τρίτου του φτωχού πληθυσμού είναι Ρωμά. Δεν είναι λοιπόν, καταλαβαίνετε την περιθωριοποίησή τους. Επίσης όσον αφορά τον ε, ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων, την κλειτοριδοεκτομή, ε, το συζητήσαμε και είναι βεβαίως πολύ σοβαρό και Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να τονίσουμε είναι η υποχρεωτική στήρωση γυναικών Ρωμά σε όλη την Ευρώπη. Οι τελευταίες περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν ήταν του 2004. Όμως έχουμε ακούσει ακόμα παράπονα που ισχύουν τώρα τα τελευταία χρόνια για τον, την υποχρεωτική στήρωση γυναικών Ρωμά και θα θέλαμε να γίνει μια έρευνα να διαπιστώσουμε τι γίνεται, αν αυτό είναι αλήθεια και σε ποια διάσταση. Ευχαριστούμε. Επόμενη μιλήτρια κυρία Μπλινκεβίτσε. Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που διοργανώσατε αυτή την ε, συνάντηση σήμερα. Και κυρίως που δώσατε τον, την ευκαιρία και σε μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να συμμετάσχουν εδώ. Θα πρέπει να ενώσουμε πραγματικά τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε την βία. Οι πολιτικοί θύνοντες, οι διάφοροι, τα διάφορα θεσμικά όργανα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Διότι αν ο καθένας δρά μόνος του, δεν θα πετύχει ο αγώνας κατά της βίας. Μας είπε ο κύριος Καρμπόφσκι ότι το κράτος μόνο του δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της βίας. Σημείωσα ότι το κράτος δεν επιτρέπεται να δηλώνει σε αδυναμία να πράξει κάτι τέτοιο. Και ποια είναι εδώ η αλήθεια. πολλά διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν από κράτο σε κράτο στην Ευρώπη των 27. Όμω το ζήτημα είναι, υπάρχουν εμπειρογνώμονε που θα μπορούσαν να εντοπίσουν διάφορε μορφέ βία. Όχι, δεν υπάρχουν αρκετοί εμπειρογνώμονε εδώ. Υπάρχει προστασία των θυμάτων. Όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Και πολλοί θεσμοί λένε ότι δεν διαθέτουν τους επαρκείς οικονομικούς πόρους. Όμως όσοι διαπράττουν την βία τιμωρούνται έστω όπως τους αξίζει. Όχι, ούτε αυτό δεν συμβαίνει. Εδώ λοιπόν θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρμπόφσκι. Πολλές φορές ακούμε την εξήγηση ότι το πρόβλημα είναι οικογενειακό, αφορά το συγκεκριμένο νοικοκυριό και πρέπει να το λύσουν μεταξύ τους. Στη χώρα μου συζητάμε εδώ και χρόνια για ένα νόμο που να καλύπτει τις περιπτώσεις οικογενειακής βίας. Δεν έχει εγκριθεί ακόμη τέτοιο νόμος, διότι κάποιοι πολιτικοί δεν κατανοούν τι θα πει η οικογενειακή βία. Για αυτούς δεν αποτελεί καν πρόβλημα. Η κοινωνία λοιπόν, η ίδια κοινωνία δυστυχώς ακόμη ανέχεται τη βία. Μια γυναίκα που είναι θύμα κάποιες μορφή βία και πάει σε κάποιο μέσο μαζική ενημέρωση και πει Δεν αντέχω άλλο, με τρομοκρατεί συνεχώ ο σύντροφό μου. Τι να κάνω, θα τη απαντήσουν, ε? Τι θε και παραπονιέσαι. Ο σύζυγό σου φέρνει λεφτά στο σπίτι. Εσύ παραπονιέσαι. Άρα η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, ανέχεται τη βία. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή, τον 21ο αιώνα. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσω με τον βούλγαρο δημοσιογράφο εδώ. Κάποιες φορές φαίνεται μάταιος αγώνας του κράτους κατά της βίας. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε άμεση δράση, διότι τα λόγια δεν φτάνουν πια, όπως είπε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Να συμφωνήσω λοιπόν εδώ με τους ευρωβουλευτές που μας είπαν ότι πρέπει να σκεφτούμε ενδεχομένως την προοπτική μιας οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και μάλιστα ήδη από φέτος. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Επόμενη μελήτρια από το Κοινοβούλιο της Κροατίας, η κυρία Γεννάκοβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της κρατικής αντιπροσωπείας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην σημερινή συζήτηση. Συμφωνούμε όλες και όλοι ότι με την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να αναλάβουμε μια διαδικασία που προαπαιτεί την πολιτική βούληση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό κατάλληλο. Στην Κροατία κάναμε αυτό το πρώτο βήμα. Δηλαδή, τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας τελευταία πέντε χρόνια εγκρίθηκαν μια σειρά στρατηγικέ, αλλά και νομοθετικέ πράξει για την προστασία κατά τη βία στο σπίτι εθνική στρατηγική ούτω ώστε να υπάρξει ισότητα των φύλων ε, μέτρα για αρρωγή και προστασία κατά τη οικογένειακή βία, ένα πρωτόκολλο για την εκδίκαση των υποθέσεων οικογενειακής βία. Επίσης, έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά την εφαρμογή των διεθνών συνθήκων. Σε συνέχεια της κύρωσής τους. Όμως η νομοθεσία δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της βίας. Χρειάζεται μακρόπνες προσπάθειες. Χρειάζεται αυτό να γίνει από πολλές πλευρές και πολλά θεσμικά όργανα σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας. Χρειάζεται μεταρρύθμιση του δικαίου. Ε, χρειάζεται ασφάλεια, χρειάζεται ε, πρόσφαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετοχή των υπηρεσιών της ε, δημοσίας υγείας. Έχουμε σημειώσει πάντως πρόοδο σε όλους αυτούς τους τομείς. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να σας πούμε ότι ακόμα απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Πέραν αυτών των βελτιώσεων έχουμε κάποια πρόοδο και όσον αφορά την ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση του κόσμου για το πρόβλημα της ε, βίας στο σπίτι, στην οικογένεια. Έχουμε συμμετάσχει στην προσπάθεια της Εκσταδίας Βουλή της Ευρώπης, στην ε, καμπάνια την διακοινοβουλευτική κατά της βίας κατά γυναικών. Πέρσι η κοινοβουλευτική μας Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων οργάνωσε μια συζήτηση στον κυρίε τραπέζι στο Κοινοβούλιο για τα προβλήματα των ε, θυμάτων της βίας όταν απεχώρησαν από τα άσυλα, από τα θεσμικά όργανα που τους βοηθούν. Θα πρέπει επομένω να προστατεύσουμε, να βελτιώσουμε την ε, ε, ζωή τους στέγαση, μόλις φεύγουν από αυτά τα καταφύγια, από αυτά τα τους οίκους προστασίας. Ε, χρειάζονται κάποια ειδικά μέτρα ούτως ώστε να τους παρασχεθεί και η ευκαιρία απασχόλησης. Και έχουμε ένα τέτοιο φορέα. Θα πρέπει να προσέξουμε τις προκαταλήψεις των εργοδοτών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ικανών πόρων γιατί θα πρέπει μπορούν να βοηθηθούν και να βρουν δουλειά τα θύματα αυτού του φαινομένου. Έχουμε επομένως ε, κάποια επιτέγματα ε, και με την ε, νομοθεσία έχουμε και μια νέα κατηγορία βίας που ονομάζεται οικονομική βία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο ιδίω στις οικογένειες με χαμηλές αποδοχές αλλά και εδώ έχει γίνει πρόοδος και σε σχέση με τα θύματα των ε, βιασμών. Και είναι υποχρεωτική πλέον η ψυχοθεραπεία των ε, βιαστών με αποτελέσματα θετικά. Φυσικά και η αντιμετώπιση της βίας είναι μακρόπνη προσπάθεια, αλλά όσον αφορά τη χώρα μας, εμείς δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας θα καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια είναι δυνατή για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιάκοβιτς. Επόμενος ε, μιλητής είναι Ευρωβουλευτής, κυρία Σουμέμπεσφέλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώ με τη συνάδελφο που εκπροσωπεί τις ε, κακομένες γυναίκες δεν είναι μόνη της. Ευχαριστούμε για την σημερινή διοργάνωση. Τώρα τα θύματα της βίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτή είναι η θέση που αρμόζει και όχι η ταπείνωση όχι η περιφρόνηση όπως γίνεται πάρα πολλές φορές και που τελικά βγαίνει κερδισμένος ο Δήμιος και όχι το θύμα. Ο θήτης και όχι το θύμα. Πολλές φορές δεν έχουμε καταγγελίες γιατί οι γυναίκες είναι απελπισμένες, είναι φοβισμένες. Εγώ είμαι θύμα τρομοκρατίας, όχι της βίας μεταξύ των ε, φίλων, αλλά ξέρω τι πάει να πει βία και θα αναλάβω ως Ευρωβουλευτής μια σχετική έκθεση. Ελπίζω αυτό να είναι χρήσιμο και ελπίζω τελικά αυτό να αξιοποιηθεί και από τα 27 κράτη-μέλη, να προστατεύσει και τις γυναίκες και όλους όσους γενικότερα χρήζουν προστασίας. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στην πολιτική μας. Θα πρέπει η καλή ιδέα να παγιωθεί με σωστές ενέργειες. Μέσα από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Γυναικών, την Επιτροπή ε, Δημοκρατικών Δικαιωμάτων θα πρέπει επομένω οι πιο αδύνατοι να έχουν στα χέρια τους κάτι που να τους προστατεύει. Να μην είναι κενό γράμμα. Να μην μείνουμε μόνο στους τίτλους των πρωτοσέλιδων όπου μέσα σε μια μέρα ξεχνιέται το θύμα. Το θύμα όμως το ίδιο δεν ξεχνάει ποτέ, ούτε εγώ θα ξεχάσω ποτέ. Και γι' αυτό και νιώθω ελέγγυα με όποιον υποφέρει. Σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα για τα θύματα. Γιατί πολλές φορές είναι, είναι φημωμένα τα θύματα γιατί αυτός που άσκει τη βία ταυτόχρονα φημώνει το θύμα του. Άρα να τους δώσουμε τη φωνή που χρειάζονται ούτως ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν, να ακουστεί η φωνή τους. Ευχαριστώ πολύ και από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο είναι η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Καρνέιρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οπωσδήποτε βλέπουμε βίες συμπεριφορές να υπάρχουν ακόμη και σήμερα και μιλάμε για ενέργειες κατά της ανθρωπότητας. τα φαινόμενα αυτά γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο και μιλάμε για μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τρόπο πολύ συγκεκριμένο που πλήττει την αξιοπρέπεια των γυναικών. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω και δεν πρέπει να σταματήσουμε και εμείς να το επαναλαμβάνουμε διαρκώς μέχρι να εξεύρουμε τρόπους να, να καταπολεμήσουμε τέτοια φαινόμενα που συστηματικά επαναλαμβάνονται. Ήθελα να κάνω κι εγώ μια-δυο παρατηρήσεις σε σχέση με τις λύσεις που έχουν βρεθεί στη χώρα μου για τα θέματα αυτά. Η Πορτογαλία, όπω και οι περισσότερε χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία για την καταπολέμηση της οικογένειακή βίας και ήταν ε, πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τρία που ελήφθησαν ε, για την με την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα με τυποποίηση των νομικών μέτρων ε, δόθηκε ορισμός για την βία κατά των γυναικών στον ποινικό κώδικα. Προέκυψε λοιπόν εντατικοποίηση το, της τιμωρίας των δραστών, της επιβολής ποινών και δεν μιλάμε πλέον ε, μόνο για θύματα αλλά και για αυτούργους, για δράστες. Βεβαίω δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ορολογία του θύματο εδώ και απευθύνομαι εδώ στην Ευρωβουλευτή που το ανέπτυξε το σημείο αυτό. Δεν γίνεται στην νομική ορολογία και την ερμηνεία που μα απασχολεί να αποφύγουμε τον όρο θύμα. Επίση, θέλαμε να καλύψουμε έναν αριθμό όσο δυνατόν μεγαλύτερο του πληθυσμού για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση και γι' αυτό διευρύναμε το δίκτυο των ε, δομών που προσφέρουν στήριξη στα θύματα και τα παιδιά τους, κέντρα στήριξης λοιπόν των γυναικών που είναι θύματα βίας και επίσης έγιναν και εξτατείς ενημέρωσης για τους αστυνομικούς που ασχολούνται ακριβώς με τα θύματα συγκεκριμένων μορφών βίας ή εκστρατείας μικτές ε, ενημέρωσης της νεολαίας, πώς προληπτικά να ετοιμαστούν οι νέοι για να μην αναπαράγουν πρότυπα βίας συμπεριφοράς. Επίσης, επιτρέψτε μου να συνεχίσω, ότι η στήριξη των θυμάτων ε, ε, ενδυναμώθηκε με, μια, με ένα νόμο που εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα για να καταπολεμηθεί ακόμη πιο εντατικά η βία κατά των γυναικών. Να προσθέσω εδώ σε σχέση με όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν προηγουμένως στη συζήτηση για τα διάφορα μέτρα για την ανάγκη εναρμόνισης, για τις μορφές παρέμβασης στις διάφορες χώρες της Ευρώπης, για το πώς πρέπει να καλύπτουμε ένα φάσμα φαινομένων, να είναι πιο συνολική προσέγγιση και ορισμός της βίας κατά των γυναικών. Ωστόσο, μεταξύ, να προσθέσω μια παρατήρηση γενικού χαρακτήρα. Το εξής. Στις περισσότερες από τις χώρες μας έχουμε και μια σημαντική βελτίωση της διαβίωσης ε, του πληθυσμού. Όμως κάποια μέρη του πληθυσμού παραμένουν ευάλωτα. Και αυτό κατακαιρματίζει και υπονομεύει τη γενικότερη αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Και υπάρχουν και άλλα φαινόμενα που μας οδηγούν ε, να προβληματιζόμαστε αυξάνεται και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Άρα τα, οι πολίτες έχουν περισσότερα προσόντα και θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν με καλύτερο τρόπο την βία. Όμως, αντί να μειώνονται τα φαινόμενα βίας, αυξάνονται, τα αντικοποιούνται και ιδίως στις ομάδες των νέων. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Σε άτομα που βρίσκονται στη σχολική ηλικία και δεν θα έπρεπε να παρουσιάζουν τέτοιες μορφές συμπεριφοράς. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες όλο και πιο συστηματικά συμμετέχουν στον αγορά απασχόλησης και στην παραγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων. Όμως αυτό από την άλλη φέρνει μορφές συμπεριφοράς που όπως βλέπουμε η βία παραμένει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει τέτοια συνολική νομοθετική κάλυψη, τέτοια ευρεία προσέγγιση και για, για τον εντοπισμό, τον ορισμό, την κατηγοριοποίηση, την επιβολή ποινών, για τις παρεμβάσεις μας, διότι τα θύματα δεν παρακολουθούνται επαρκώς. Είναι πολλές φορές θύματα της κακής υλοποίησης των υπευθύνων για τους νόμους. Αυτό συνεχίζεται και λόγω της διαρκούς παρουσίας στερεοτύπων προκαταλήψεων και από άποψη κοινωνική και πολιτιστική και νομοθετική, αυτό είναι ένα θέμα, μια συμπεριφορά που πρέπει να καταπολεμηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι να ε, ευαισθητοποιηθούμε, να κινητοποιηθούμε και ιδίως οι πολιτικοί ηθήνοντες να ενισχύσουν τους πολιτικούς και νομοθετικούς μηχανισμούς. Διότι πιστεύω εδώ θα πρέπει να έχουμε ακόμη και συμμετοχή των κοινοτήτων θα πρέπει οι ίδιες οι κοινότητες πολιτών να αναλάβουν ευθύνες για να υποδεχτούν και να στηρίξουν θύματα που ενδεχομένως ζουν στο πλαίσιο τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέτμαν ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που επιτέλους μιλάμε για το θέμα αυτό της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Ε, στη χώρα μου μέχρι πριν από 15 χρόνια ήταν θέμα ταμπού. Δεν ακουγόταν αν μια γυναίκα ε, κατήγγειλε τον άντρα της ότι την έδρανε. Τότε της έλεγαν οι αρχές αποκλείεται. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Ε, αυτά που λες είναι ψέματα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που συζητούμε αυτό το, το, θέμα διότι η βία παρουσιάζεται παντού και στο σπίτι και στα σχολεία και στην ε, δημόσια ζωή. Πιστεύω ότι αυτή, αυτός ο οργανισμός, το Ίδρυμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια θαυμάσια διοργάνωση και θα πρέπει να ζητήσει από τα εθνικά κοινοβούλια να σεβαστούν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην ε, χώρα μου υπάρχουν βεβαίως σπίτια προστασίας για τις γυναίκες αλλά και για τα παιδιά που είναι ένα θαυμάσιο δίκτυο προστασίας και καταφυγίου. Είναι τα σπίτια καταφύγια. Αυτά λοιπόν τα κάτι καταφύγια όπου οι γυναίκες και τα παιδιά μπορούν να, να καταφύγουν για να μείνουν και να αποφύγουν να, γίνουν... να συνεχίσουν να είναι σήματα βίας πρέπει να καλύπτονται από ένα νομικό πλαίσιο και πρέπει να, να... να δημιουργηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκοερέιδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Όχι μόνο λόγω των συνεισφορών που συγκεντρώσαμε από διαφορετικές χώρες, αλλά και γιατί τα θέματα που αναπτύσσουμε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ξέρουμε ότι τα ζητήματα τα σχετικά με την βία είναι σοβαρά και μπορεί να έχουν να κάνουν από την εμπορία ανθρώπων και παρόλο που ζούμε σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, ξέρουμε ότι ετησίως 15.000 γυναίκες είναι θύματα διακίνησης, εμπορίας. Και στο συντριπτικό τους ποσοστό για σκοπούς ε, εκπόρνευσης ή παράνομης εργασίας, πολλές από αυτές είναι από τις χώρες μας και είναι θύματα συνθήκων διαβίωσης ε, προσωρινής ευτόχειας μάλλον ή προσωρινής εργασίας. Και είναι και θύματα δικτύων ε, της παραοικονομίας, της μαφίας που πολλές φορές τις οδηγούν σε τρίτες χώρες. Η σκοπή είναι πάντοτε η ίδια, η εκμετάλλευση η υποβάθμιση του, της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Όμως οι ρίζες του προβλήματος είναι πάντοτε η ίδια. Φτώχεια, εκμετάλλευση, ανισότητα. Θα πρέπει Λοιπόν, να δούμε τι δράση θα αναλάβουμε σε διάφορα επίπεδα. Δεν αρκεί να έχουμε ένα παρατηρητήριο. Σημαντικό είναι και αυτό. Και η τηλεφωνική γραμμή καλή είναι. Όμω, είναι αναγκαίο να πάμε παραπέρα Χρειάζονται νόμοι οι οποίοι να καταστέλουν, να αναχαιτίζουν αυτού του είδους την εμπορία και να λαμβάνουν δραστικά μέτρα κατά των δικτύων της μαφίας. Θα πρέπει να στηρίξουμε επίσης τα θύματα. Θα πρέπει να εργαστούμε στον τομέα της πρόληψης, δηλαδή να επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια του προβλήματος, να εξασφαλίσουμε στις γυναίκες οικονομική ανεξαρτησία, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσουμε τη βία. Προφανώς υπάρχει και η βία στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό σε όλα τα κρατημέλη ισχύει. Πολλά από τα θύματα αυτής της οικογενειακής βίας σε κάθε μια από τις χώρες μας πρέπει να μας θυμίζει ότι πέραν της επιβολής ποινών στους δράστες, την εντοπισμό των φαινομένων βίας, πρέπει να καλύψουμε και να στηρίξουμε τα θύματα, να εξασφαλίσουμε την άσκηση όλων των, δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων τους, την αξιοπρεπή διαβίωση, να τους δώσουμε δυνατότητες να ξεφύγουν από τη βία, όχι να παραμείνουν εχμαλωτισμένες. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εκστρατείες ενημέρωσης για την ισότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συμμετοχή που μπορεί να έχουμε στις χώρες μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τους κρατικούς οργανισμούς, τις ενώσεις και συλλόγους των πολιτών και γυναικών. Όλες αυτές οι συνεισφορές θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Είναι πολλαπλές οι δράσεις που μπορούν να αναλυφθούν και οι πολιτικοί θυνόντες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνε τους, το σημαντικότερο μέρος αυτή της δράσης και σε αυτήν την φάση προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε, να προβάλλουμε τις πτυχές αυτών των φαινομένων και να απαιτήσουμε τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κολέ Ντιουτρόι από το Ευρωπαϊκό Γυναικείο Λόμπι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών, να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μας για τη συζήτηση που γίνεται εδώ και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση είναι κάτι που είναι ένα κοινό στοιχείο σε όλη την Ευρώπη αυτό και σε όλο τον κόσμο βεβαίω. Και απασχολεί πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Το δικό μα δίκτυο εκπροσωπεί οργανώσει γυναικών σε όλα τα κράτη τη Ευρώπη και τι χώρε τι ε, προενταξιακέ. Εδώ και χρόνια λοιπόν όχι μόνο να αποδείξαμε τη σημασία και επιβάλαμε την αναγνώριση του φαινομένου αυτού, δηλαδή του γενικού χαρακτήρα που έχει η ανδρική βία κατά των γυναικών, αλλά εντοπίσαμε και τις μορφές βίας. Και όχι μόνο συζητήσαμε εδώ διαμακρών αυτές τις μορφές, αλλά και τις αιτίες, την ανισότητα ανδρών γυναικών δηλαδή, την σημασία που έχει να αντιμετωπιστεί εξάπλωση αυτού του φαινομένου και να το δούμε και από μια άλλη προοπτική. Αυτή η προοπτική σήμερα είναι διτή. Να συζητήσουμε βεβαίω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί εδώ και χρόνια ζητάμε μια οδηγία για μια σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική που να εξασφαλίζει ισότιμη προστασία στις γυναίκες, την ίδια πρόληψη. Μια πολιτική που να διασφαλίζει ότι και οι άνδρες θα κατανοήσουν περί ο λόγος. Και έπειτα, η δεύτερη πτυχή είναι ότι σήμερα βλέπουμε την βία των ανδρών κατά των γυναικών να αρχίζει να θεωρείται μορφή διάκρισης και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ήδη λέγεται και ήδη αναφέρεται στα διεθνή κείμενα από το Πεκίνο, από τις συναντήσεις κορυφής που ήδη έχουμε συζητήσει εδώ με τις ε, συμβάσεις του ΟΗΕ κατά όλων των διακρίσεων. Τώρα έχουμε τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ανάλογη χάρτα Εκεί αναφέρεται ρητό ότι δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά τέτοια φαινόμενα ανδρική βία κατά των γυναικών. Δεν μπορεί να είναι τόσο διαδεδομένα. Δεν μπορεί να, έχει, να λαμβάνουν τόσο λίγη μέρημνα τα κράτη-μέλη για τέτοια θέματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Για το θέμα των εμπειρογνωμόνων και για να απαντήσω εδώ σε μια προηγούμενη παρέμβαση, εμπειρογνώμονε υπάρχουν έχουν περάσει και από εδώ και πολλοί συνάδελφοι θα μπορούσαν να το σχολιάσουν αυτό. Υπάρχουν και κυβερνητικέ οργανώσει γυναικών που εργάζονται από χρόνια στην ε, πραγματική καθημερινή ζωή. Κάποιε φορέ στερημένε και από τα απαραίτητα μέσα. Κάποιε φορέ υποδεχόμενε και φιλοξενώντα ε, στα διαμερίσματα των μελών γυναίκε θύματα. Υπάρχουν αυτά και η εμπειρογνωμοσύνη μας έχει χτιστεί μέρα με τη μέρα και με την άσκηση πίεσης που κάνουμε εδώ και χρόνια πετύχαμε ένα παρατηρητήριο να, δι... ιδρυθεί ένα παρατηρητήριο, ένα παρατηρητήριο που βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από όλα όσα ακούσαμε σήμερα υπάρχει συνεχώς αυτή η διαρκής αναζήτηση του αυγού και της κότας. Αναρωτιόμαστε δηλαδή το μόνο πρόβλημα είναι οι υπηρεσίε που θα προσφέρουμε στι γυναίκε, η μέρημνα και το δικαίωμα να τι επιτρέψουμε να μιλήσουν ή τα στατιστικά στοιχεία που θα αποδείξουν την σοβαρότητα του προβλήματο. Οι πολιτικοί που σήμερα βρίσκονται μεταξύ μας, οι βουλευτές, θα πρέπει να προωθήσουν καλύτερα νομοθετικά μέτρα. Την ανάληψη δηλαδή δράσης και νομίζω ότι και οι δύο ενέργειε πρέπει να αναλυθούν παράλληλα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω ταυτόχρονα και εσάς για την πρωτοβουλία σας, αλλά και όλους τους συναδέλφους που μοιράστηκαν μαζί, τους, μαζί μας τις εμπειρίες τους. Πολιτικές εμπειρίες, θεσμικές, θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Άνια από τη Σουηδία είναι η επόμενη ομιλήτρια, πρόεδρος της, του Σουηδικού Οργανισμού για τις Γυναίκες και τις Νέες Γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε, σε, αυτήν, ε, την, ε, σε αυτό το συνέδριο, σε αυτή την ακρόαση και θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους χαιρετισμούς όλων των γυναικείων οργανώσεων στη Σουηδία. Και θα δώσουμε μάλιστα και ένα βραβείο στην εκπρόσωπό μας η οποία ανακηρύχθηκε η γυναίκα ε, του έτους ε, στη Σουηδία. Η Σουηδία ήταν πάρα πολύ δραστήρια στο γυναικείο κίνημα και έχει προχωρήσει πάρα πολύ η σουηδική νομοθεσία. Ε, αυτό το οφείλουμε σε μεγάλο ποσοστό στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιστεύω ότι έχουν εργαστεί θαυμάσια προς τους κοινού μας στόχους και υπάρχουν τώρα, υπάρχει μια πληθώρα νομοθεσίας για το θέμα των γυναικών. Το, κοινοβούλιο, το Εθνικό Κοινοβούλιο στη Σουηδία ε, ακούει πολύ προσεκτικά όσα λέγονται από τις γυναικείες οργανώσεις και έχουμε ένα, μια δέσμη μέτρων ε, υπέρ των γυναικών ε, για την οποία είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Το πρόβλημα στη Σουηδία περισσότερο αφορά την πλευρά της εφαρμογής, της υλοποίησης. Εάν ε, δεν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους νόμους, μπορούν οι νόμοι αυτοί να είναι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά ποιο θα είναι το νόημα δεν εφαρμόζονται. Τα έργα λοιπόν πρέπει να γίνουν πράξεις. Επίσης πρέπει να συνεργαστούμε στενά και να ακούσουμε τη φωνή των ε, ε, γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν περάσει από αυτή την ε, ε, φρικτή εμπειρία της βίας εναντίον τους και, και στο σπίτι και σε άλλους χώρους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθω εδώ πιστεύω ότι θα έχει υλοποιηθεί η εφαρμογή των νομικών μέσων που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Πολύ την Άντζελα Μπουσό. Αυτή ήταν η τελευταία μελήτρια και θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, ε τρεις ε, καλεσμένους μας στο πάνελ για να ε, ολοκληρώσουν και για να πούν μερικά λόγια συμπερασματικά για τη συνεδρίασή μας αυτή. κυρία Αλμπέρντι. Ε, ε, μικρόφωνο παρακαλώ, δεν ακούγεται η ομιλήτρια. Μικρόφωνο παρακαλώ. Διαπιστώθηκε σήμερα ότι υπάρχει προβληματισμός και αλλά έχει τεθεί και ένας κοινός στόχος η καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών. Σε όλες τις παρεμβάσεις τονίστηκε κάθε θέμα που μας ε, απασχολεί, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη, προστασία, αρρωγή κατά θυμάτων και κυρώσεις κατά των εγκληματιών. Επομένως, σε όλες τις ε, χώρες θα πρέπει να γίνει ένα συντονισμός να ενώσουμε τις προσπάθειές μας να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να υπάρξει κάποιο είδους αμοιβαία αρρωγή. ότι και στον ΟΗΕ δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση και χρειαζόμαστε την βοήθεια της Ευρώπης. Υπάρχουν δε δύο πάρα πολύ σημαντικές ε, ε, πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Πρώτα πρώτα είναι αυτή η εκστρατεία ε, ενωμένη εναντίον της βίας, αυτή η εκστρατεία του Γενικού Γραμματέα που το αρμόδιο όργανο του ΙΕ έχει αγκαλιάσει και προσπαθεί να υλοποιήσει την προσπάθεια αυτή σε σχέση με την οποία από πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εμπλακεί και οπότε παρακαλώ συνεχίστε προς την ίδια κατεύθυνση καταβάλλετε και στο μέλλον αυτές τις προσπάθειες να διαδοθεί αυτή η εκστρατεία να τονιστεί το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε ε, κυβερνήσεις με κυβερνητικές οργανώσεις, ε, φορείς, ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όσο περισσότερο ενώνουν τις προσπάθειές μας, τόσο περισσότερο θα καταφέρουμε να αλλάξουν νοοτροπίες και να εκριζώσουμε, να σταματήσουμε αυτή την βία. Υπάρχει μια δεύτερη πρωτοβουλία για την οποία σας μίλησα. Ήταν αυτό το, το Ταμείο Ίδρυμα για χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί η βία. Και αυτό το ταμείο χρειάζεται όμως πόρους. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πάρα πολύ γενναιόδρες όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Οπότε παρακαλώ ε, βοηθήστε ούτως ώστε να υπάρξει επιρροή προς αυτή την κατεύθυνση και ούτως ώστε με πόρους ε, οικονομικούς να βοηθηθεί αυτό το ταμείο του ΟΗΕ να έχει μηχανισμούς και συγκεκριμένα προγράμματα για την καταπολέμηση της ε, βίας παντού στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αλμπέρτη. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ακούσουμε όμως τον κύριο Καμπόφσκι στα τελευταία του σχόλια. Κοιτάξτε, πριν από λίγο τέθηκε το ζήτημα της, των αιτιών της βίας κατά των γυναικών και παιδιά γενικά. Η απάντηση είναι απλή και είναι η εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν τη βία το κάνουν επειδή τους επιτρέπεται επειδή είναι ελεύθεροι να το κάνουν και επειδή οι εθνικές ε, υπηρεσίες και φορείς δεν παρεμβαίνουν. Το κράτος πρέπει να εξανθρωπίσει αυτά τα άτομα. Η Ευρώπη δεν είναι αρκετά θαραλέα όταν ερχόμαστε στο θέμα της βίας, ε, στις, ε, ας πούμε, πολιτισμικές παραδόσεις ε, μειονοτικών εθνοτήτων ε, ή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ πιο θαραλέα και αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Εν κατακλείδη ήθελα να πω ότι δεν θα ήθελα οι γυναίκες από τη δική μου χώρα να μεταναστεύσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορέσουν να ζήσουν με ασφάλεια και με ελευθερία και να απαλλαγούν από τον τρόμο αυτό της βίας. Εάν αυτό συμβεί τότε θα είναι οι μετανάστριες ε, για πολιτικούς. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μόρτον ε, Κάουιλ. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάτσι έθιξε το θέμα της συλλογή στοιχείων αλλά και της μελέτης των στοιχείων και τι υποκρύπτεται πίσω από αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η μελέτη που σας είπα, η MIDIS, η EU MIDIS, η οποία αφορούσε τις ε, μειονότητες, εθνότητες και ε, ε, ειδικέ ομάδες, είχε ως στόχο την καταγραφή πληροφοριών για να μπορέσουμε να με τη μελετήσουμε και για να συνάγουμε συμπεράσματα. 23.500 άτομα ε, έδωσαν στοιχεία και Ρωτήσαμε το ποσοστό των, γενικό, γυναικών, πολύ υψηλό, 27% που μας είπε ότι είναι σήματα βίας, ε, αν το κατήγγυλαν και όταν μας απάντησαν αρνητικά, ρωτήσαμε γιατί δεν το κατήγγυλαν. Μας είπαν λοιπόν διάφορες δικαιολογίες, πολλές από τις γυναίκες φοβόντουσαν και πολλές δεν είχαν πληροφορίες για το πού μπορούν να καταγγείλουν αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό ε, σας ε, παραπέμπω σε αυτή τη μελέτη EU Minds του, της υπηρεσίας μου, του οργανισμού μου. Δεύτερον, αυτό που ανέφερε, που ανέφερε η κυρία Στόμψον και η Γιούρικα είναι η πολλαπλή η πολλαπλή διάκριση, όχι μόνο διάκριση και ε, ε, το φαινόμενο της βίας, αλλά και άλλες διακρίσεις, παραδείγματο χάρη ψυχικές και σωματικές ε, διακρίσεις, ψυχική και σωματική βία, σε, εναντίον συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και των γυναικών μέσα σε αυτές τις ομάδες. Άρα λοιπόν αυτό το σημειώσαμε και θα το εξετάσουμε. Τις ε, ε, πολυδιάστατες διακρίσεις. Επίσης, ε, σημείωσα τη, την ε, σημασία ε, της Στοχόλμης, του, της συμφωνίας της Στοχόλμης και θα κοιτάξουμε τι πρόοδο έχει επιτευχθεί βάσει των δεσμεύσεων της Στοχόλμης και πώς θα μπορέσουμε να να προστατεύσουμε καλύτερα τα σήματα. Δεδομένου ότι, όπως είπαμε, η βία άπτεται της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε μηχανισμούς προστασίας για τα σήματα. Και ακριβώς αυτό θα μελετήσουμε για τα επόμενα χρόνια ε, το Ίδρυμα ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ε, ε, ενδιαφέροντα σχόλια και τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Μέρος της εντολής μας είναι να καταγράψουμε τις καλές πρακτικές που υπάρχουν, που έχουν εφαρμοστεί ε, για να χρησιμοποιήσουμε την ε, εμπειρία αυτή ε, για την εξέβρεση λύσεων και προτάσεων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν από τεχνικά κοινοβούλια σήμερα μαζί μας. και επίσης και τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα τώρα να κλείσω την σημερινή μας ακρόαση σημειώνοντας ότι αφού ακούσαμε όλες τις ομιλίες του σημερινού πρωινού νομίζω ότι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει ένας αριθμός ε, οργανώσεων γυναικών στην Ευρώπη που τους με ευγνωμοσύνη για το έργο τους που εργάζονται σκληρά για την προστασία των γυναικών με τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, έχουν ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη και τους πολιτικούς των εθνικών κυβερνήσεων να φέρουν αυτό το θέμα στο επίκεντρο της προσοχής τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε όλες και όλους όσους βοήθησαν και χάρη στο δικό τους έργο να έχουμε μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων μας αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να σταματήσουμε τη βία και θα τη σταματήσουμε. We can stop it. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας τη σημερινή μας ακρόαση και να σας θυμίσω ότι υπάρχει δεξίωση για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου στον δεύτερο όροφο. Απλώς κατεβείτε τις καλες μέχρι τον από κάτω όροφο και εκεί υπάρχει δεξίωση. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Και ευχαριστώ και όσους βοήθησαν για την διοργάνωση της σημερινής ημέρας, καθώς και τους διερμηνείς που έκαναν πολύ καλή δουλειά, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Γεια σας.